Ladies and gentlemen. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Καταρχήν, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δεν βλέπω παρατηρήσεις, άρα μπορούμε να την εγκρίνουμε. Θα ήθελα για την ημερήσια διάταξη να πω ότι η συζήτηση θα γίνει αύριο το πρωί για την κατάσταση στην Αίγυπτο. Παρουσία του Κριστιαν Μπέργκερ, του Διευθυντή της ΑΕΔ Και δεύτερον, θα ήθελα να προσθέσουμε ένα νέο σημείο στην ημερήσια διάταξη, την ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του, κυρίου, του Μαυροβουνίου, τον κύριο Ράγκο Κρυόκαπιτς. Και αυτό θα γίνει αύριο, ημέρα Τρίτη, στις 4 το απόγευμα. Ανακοινώσεις δεν υπάρχουν εκ μέρους του Προέδρου. Next item, which is of mini... Ας περάσουμε στο τρίτο σημείο, την έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 18ης Οκτωβρίου, 25ης Οκτωβρίου, 15ης Νοεμβρίου,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 Μήπως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με την έκθεση Βάιντερ, ε? γιατί ο Σκιώδης ε, εισηγητής μας ευκαιρεί μόνο το πρωί, στην αρχή της συνεδρίασης, ε, να έρθει. Θα ήθελα να παρακαλώσω λοιπόν να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία με την έκθεση Βάιντερ, αν δεν έχετε αντιρρήσει. Ο Πρόεδρος. Να ρωτήσω τον κύριο Πρέντα, συμφωνεί για την αντιστροφή αυτή των σημείων. Κύριε Ρότσεκ, το ίδιο. Ωραία. Μια και οι συνάδελφοι δείχνουν κατανόηση, μπορούμε να τροποποιήσουμε τη σειρά των σημείων για ψηφοφόρια αύριο. Επανέρχομαι λοιπόν στην έγκριση των πρακτικών. Επαναλαμβάνω, εγκρίνουμε τα πρακτικά συνεδριάσεων της 18 η Οκτωβρίου, 25 25η Οκτωβρίου, 15ης Νοεμβρίου και 26 η και 27 η Νοεμβρίου 2012. Αν δεν υποβληθούν ε, αστάσεις και αντιρρήσεις θα θεωρήσουμε ε, ως εγκεκριμένα τα πρακτικά. Σημείο 4 τώρα της ημερήσης διάταξη. Συνολική έκθεση παρακολούθησης ε, του 2012 για την Κροατία. Πριν ε, περάσουμε στη δεύτερη συζήτηση του σχεδίου έκθεση για την Κροατία, θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότατα μία αντιπροσωπεία μελών της Κρατικής Βουλής που πραγματοποιούν ε, επίσκεψη ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αγαπητοί φίλοι, η... τιμάτε ιδιαίτερα ε, με την παρουσία σας την Επιτροπή μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν, ως ευχαρέστητε. Ντόμπρο Ντόσλι. So, let us now turn to... Και επανερχόμαστε στο θέμα της σας διάταξης, το 4, την ε, εξέταση του σχεδίου πρώτες ψηφίσματος, που θα είναι το τελευταίο που θα υποβάλει η Επιτροπή μας για την Κροατία. Η Κροατία θα γίνει το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουλίου του 2013, το τρέχοντος έτους. Μέχρι στιγμής 24 ε, κράτη-μέλη και η Κροατία έχουν εγκρίνει την ενταξιακή συνθήκη έχουν κυρώσει την ε, ενταξιακή συνθήκη και θα ήθελα επ' ευκαιρία να απευθύνω έκκληση προς τα κράτη-μέλη που δεν έχουν κυρώσει ακόμη τη συνθήκη αυτή, ε, την Γερμανία, τη Δανία και την Σλοβενία, να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κύρωσης της ενταξιακής συνθήκης της Κροατίας και μάλιστα εμπρόθεσμα, ώστε να προλάβει αυτή η χώρα να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τηρώντας το ομόφωνα εγκριθέν χρονοδιάγραμμα γι' αυτό. Επίσης ε, χαιρετίζω τις προσπάθειες ε, των κυβερνήσεων της Κροατίας και της Σλοβενίας προκειμένου να αναβρεθεί ε, λύση στην υπόθεση της τράπεζας της Λιουμπλιάνα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας τον κύριο Ρόουτζεκ για να μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση των 62 τροπολογιών και των 5 συμβαστικών τροπολογιών για την έκθεση αυτή παρακολούθηση Κροατίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς πρόκειται για τη δεύτερη εξέταση. 62 τροπολογίες ε, κατατέθηκαν, οι περισσότερες είναι πολύ επικοδομητικές και ευθυγραμμίζονται με τα συμπεράσματα της έκθεσης μας. Η κατάρτιση της έκθεσης και η προετοιμασία της έδειξε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ενωμένο και συσπηρωμένο και υπάρχει μια διακομματική συμφωνία που λέει ότι η Κροατία βρίσκεται σε καλό δρόμο και θα προσχωρήσει την πρώτη η Εβδόμου του 2013. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρώσει τα 10 καθήκοντα που της έχουν απομείνει και από την τελευταία επιτροπή και οι, οι τελευταίες υποχρεώσεις είναι οι, οι εργασίες που θα γίνουν στο διάδρομο Νόιν στην Αδριατική θάλασσα θα ολοκληρωθούν τον Απρίλιο. Οι περισσότερε τροπολογίε αφορούν το μακροπρόθεσμο στόχο της κροατία, δηλαδή ενίσχυση της δικαστική εξουσίας, ε, της επιβολής του κράτου δικαίου και την πάταξη της διαφθοράς ιδιαίτερα σε υψηλά κλιμάκια. Επίσης, ε, θα πρέπει η αποκατάσταση του κράτου δικαίου να αποτελεί προτεραιότητα της, κυβερνή, της ε, όχι μόνο μέχρι την ένταξη, αλλά και μετά, γιατί πρόκειται για μια ε, δυναμική διαδικασία που βρίσκεται εν εξελίξη δηλαδή. Και άλλωστε υπάρχει και διακομματική συμφωνία στην Κροατία. Γι' αυτό έχουμε και αντιπροσωπεία από την Κροατική Βουλή, το ΣΑΜΠΟΡ και από εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών. Οι συμβαστικέ τροπολογίε αφορούν τον περιφερειακό ρόλο τη Κροατία για την περαιτέρω σταθεροποίηση και διεύρυνση στην περιοχή και απευθύνουμε έκκληση προκειμένου να διευθετηθούν οι διμερείς ε, διαφορές και να μην δημιουργήσουν προσκόμματα στις ε, ενταξιακές διαδικασίες των γειτονικών χωρών. Έχει μείνει ακόμη κρεμέ στο θέμα της Λιουμπλιάνσκα Μπάνκα, της τράπεζας ε, της Λιουμπλιάνα. Είχαμε μια συμφωνία των πρωθυπουργών που κατέληξαν σε μια άτυπη συμφωνία και στις 11 Μαρτίου θα έχουμε επίσημη συνάντηση των Πρωθυπουργών της χώρας μετά τη Συμφωνία των Υπουργών Εξωτερικών και ελπίζω να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Άλλωστε και οι δύο πλευρές έχουν επίγνωση της σοβαρότητας της κατάστασης και της ανάγκης να βρεθεί κατεβηγόντως μία λύση μέχρι το Μάρτιο δηλαδή να καταλήξουν οι Πρωθυπουργοί σε μια συμφωνία που θα γίνει δεκτή και από τις κυβερνήσεις και από τα κοινοβούλια. Είναι σημαντικό αυτό και για την Σλοβενική Βουλή για να προχωρήσει και στην κύρωση τη ε, δεξιακή συνθήκη τη Κροατία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και του σκιώδει μα ηγητέ για την πολύ επικοδομητική του ε, συμβολή. Υπάρχει συνένεση, όπω σα είπα, και περιμένω να ακούσω τα σχόλιά σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε εισηγητά. Θα δώσω τώρα το λόγο στους σκιώδεις μας εισηγητές, αρχής γενομένης από τον κύριο Μπέρν Πόσελτ. Ζητώ συγγνώμη καταρχήν γιατί είμαι κάπως ε, κρυωμένος και γι' αυτό ακούγεται έτσι η φωνή μου. Θα ήθελα να πω ότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά με τον κύριο Ρουτσέκ. Μπορέσαμε να φτάσουμε σε μία συνένεση μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων και φτάσαμε σε ε, απτά αποτελέσματα και θέσαμε τις βάσεις για την προσχώρηση της Κροατίας. Θα ήθελα να κάνω μία μικρή διόρθωση, γιατί η έκθεση αυτή είναι μία έκθεση για να αποφανθούμε ως προς την παρούσα κατάσταση σε σχέση με τον ε, έλεγχο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς όμως ως ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε δεσμευθεί ως προς την προσχώρηση της ε, Κροατίας την 1η Δεκεμβρίου του 2011 εμείς εγκρίναμε την προσχώρηση. Δεσμευτήκαμε δηλαδή. και μετά από το δημοψήφισμα όπου αποφάνθηκε ο κροατικός λαός. Όλοι οι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων υπέγραψαν την συνθήκη προσχώρησης. Μερικοί προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι ξανανοίγει η διαδικασία παρά την εξαιρετική έκθεση του εισηγητή του κυρίου Ρούτσεκ. Πρόκειται για έναν δεκάλογο σημείων που έχουν ενταχθεί στην έκθεση παρακολούθησης που θα υποβάλει η Κομισιόν στο εγγύς μέλλον. Γι' αυτό θα ήθελα να μην δημιουργηθεί η αντίληψη ότι εισάγονται νέα ζητήματα. Γι' αυτό το λέω προς τις τρεις χώρες οι οποίες δεν έχουν ακόμα κυρώσει. Δηλαδή τη Σλοβενία, τη Δανία και τη δική μου χώρα. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό το ότι η Γερμανία, η οποία υποκίνησε αυτή τη διαδικασία, στη συνέχεια κράτησε αυτή τη στάση, την επιφυλακτική στάση. Δηλαδή, καθυστερούμε με την κύρωση. Δεν υπάρχει πολιτικό κίνητρο γι' αυτό, όμως θεωρούμε ότι θα πρέπει να επισπεύσουμε τη διαδικασία και ας μην υπάρχει πολιτικό κίνητρο για την καθυστέρηση αυτή. Χαίρομαι λοιπόν ότι, για το γεγονός ότι καταφέραμε να πούμε ότι δίνουμε πράσινο φως για να προσχωρήσει η Κροατία την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, όπως είχε συμφωνηθεί από τις συνθήκες. Και προτρέπουμε τις χώρες που δεν έχουν κυρώσει την ε, συνθήκη προσχώρησης να το πράξουν άμεσα. Όπως ξέρετε, έχουμε Κροάτες παρατηρητές και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό πριν από τη λήξη της διαδικασίας. Ευχαριστούμε κύριε Πόσελτ. Ο Ιβο Βάιγκο έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Συμμερίζομαι αυτά που μόλις προείπε ο κύριος Πόσελτ. Εμείς δεν θέλουμε να θίξουμε νέα ζήτηματα σε σχέση με την ε, μελλοντική προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, εργαζόμαστε έτσι ώστε η Κροατία την 1η Ιουλίου να μπορέσει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και εγώ ε, δέχομαι θετικά τους ε, εκπροσώπους του Κοινοβουλίου της Κροατίας έτσι ώστε να αποσταλεί και ένα σαφές μήνυμα προς την Κροατία από την Επίτροπή μας, την ΑΦΕΤ. Θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω, να μιλήσω για την πολύ καλή συνεργασία με τον εισηγητή, τον κύριο Ρότσεκ. Έχουμε συμφωνήσει επί όλων των θεμάτων, των επιμέρους θεμάτων, όπου υπήρξαν διάφορες ε, πολιτικές προσεγγίσεις ως προς τις προτεραιότητες. Παρ' αυτά, στο τέλος καταφέραμε να φτάσουμε σε μία συνένεση ως προς ουσιώδη ζητήματα, θεμελιώδη ζητήματα και τάσσονται υπέρ της προσχώρησης της Κροατίας. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων θα ήθελα να τονίσω ότι η ομάδα μας είχε ταχθεί αναφανδών υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ένταξη της Κροατίας. Μεταξύ των τροπολογιών από τη δική μας ομάδα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο τροπολογίες. Η μία αναφέρεται στη, στο σεβασμό των μειονοτήτων, όλων των μειονοτήτων, με βάση την εθνότητα ιδιαίτερα σε σχέση με τις λεσβίες, ομοφιλόφιλους και λοιπά, δηλαδή ως προς το σεξουαλικό προσανατολισμό και επίσης θα ήθελα να ε, στυλιτεύσω την Καθολική Εκκλησία της ε, Κροατίας για τη στάση που έχει κρατήσει στο θέμα αυτό δεν συμβαδίζει με την, ε, την ελευθερία που εμείς ε, προασπίζουμε ως προς το σεξουαλικό προσανατολισμό. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις εξελίξεις και σε αυτό το τομέα και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον ε, πόλεμο, τον πόλεμο και τις μειονότητες ε, Σέρβων στην Κροατία και Τούμπαλιν. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επαναπατρισμού, κάτι το οποίο θα πρέπει να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατόν. Ως προς την ε, Λιουμπλιάνσκα Μπάνκα, προσωπικά θα πρέπει να πω ότι είμαι πεπισμένος ότι αυτό δεν θα αποτελέσει πρόσκομα για τη διεύρυνση. Πρέπει να αναφερθεί αυτό το σημείο και όλες οι πολιτικές ομάδες συμφώνησαν υπέρ της ε, κύρωσης ως πρώτη προτεραιότητα. Παρά από αυτή τη μικρή δυσκολία και την πολιτική εξέλιξη της χώρας και της δικής μου χώρας που είναι μια ε, γειτονική χώρα. Προβλέπονται εκλογές, θα δούμε ποιος θα παραμείνει στην εξουσία και ποιος όχι. Εν πάση περιπτώσει, ε, εμείς θεωρούμε την Κροατία έναν φυσικό μας σύμμαχο. Από τη δική μας πλευρά θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να προσκαλούμε τα Εθνικά Κοινοβούλια, ε, τους εκπροσώπους του συγκεκριμένου Κοινοβουλίου, της υποψήφιας χώρας και θα πρέπει να καλέσουμε και τις χώρες που δεν έχουν κυρώσει να το πράξουν το ταχύτερο δυνατόν. Να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία. Είμαι σίγουρος ότι τα κράτη-μέλη θα κυρώσουν στα προβλεπόμενα χρονικά όρια. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπραντνερ έχει το λόγο. Thank you very much. Um, and a warm. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τους ε, Κροάτες συναδέλφους. Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρούτσεκ και τους Κιώδης για την εξαιρετική συνεργασία τις τελευταίες εβδομάδες και νομίζω ότι οι συμβαστικές προτάσεις είναι απόλυτα ισορροπημένες και αποτελούν οδηγό για την Κροατία και την Κομισιόν τους ε, τελευταίους μήνες. Έχουμε υποβάλει ορισμένες τροπολογίες έτσι ώστε να ορίσουμε καλύτερα ορισμένα υπολοιπόμενα προβλήματα που αναγράφονται και στις τροπολογίες συμβιβασμού. Όπως σας είπα, θα πρέπει να επιταχυνθεί η προσπάθεια των ε, Κροατών για το κράτος δικαίου, για την καταπολέμηση της διαφθοράς, για το ρόλο της δικαιοσύνης στα εγκλήματα πολέμου και ούτω καθεξής. Είμαι πεπισμένη ότι θα προσχωρήσει η Κροατία ε, το καλοκαίρι και όλοι το προσμένουμε αυτό το γεγονός. Με χαρά. Η διαδικασία ε, κύρωσης δεν είναι κάτι το οποίο εντάσσεται μέσα σε ε, διμερείς ε, διαπραγματεύσεις ή υπηρετεί τέτοιες σκοπιμότητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει τομείς όπου υπάρχουν ζητήματα ακόμα εκκρεμή, αλλά δεν εντάσσονται σε ένα διμερές καθεστώς. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Πόσελτ και για τη δική μου χώρα και σας ε, εύχομαι να αναρώσετε τάχιστα κύριε Πόσελτ. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο τροπολογίες μας όπου προσπαθούμε να αντλήσουμε διδάγματα από τη διαδικασία προσχώρησης της Κροατίας. Η πρώτη είναι η 56, το δεύτερο τμήμα, που σχετίζεται με, τις, ε, με τους με διμερεί μάλλον καθαρά ζητήματα. Και εμείς ζητούμε έναν ε, μηχανισμό διευκόλυνσης και διαιτησίας, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις χώρες να, επιμή να επιλύσουν διμερεί ζητήματα και να μην αποτελέσουν πρόσκομα στην ενταξιακή διαδικασία. Επίσης, θεωρούμε ότι τα διμερή ζητήματα δεν θα πρέπει να αναχαιτήσουν τη διαδικασία ένταξης. Επίσης, η τροπολογία 61 ασχολείται με την κοινωνία των πολιτών μέσα στα πλαίσια της ενταξιακής διαδικασίας και γνωρίζουμε ότι το Κοινοβούλιο της Κροατίας θα ε, αντλήσει αυτά τα διδάγματα για τους ε, μελλοντικούς, ε, το μελλοντικό κύκλο διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ πολύ και τον προτέρων για την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Μόνικα Μακοβέη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω ε, την Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος και χαιρετίζω τον κροατικό λαό. Δεύτερον, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον εισηγητή, διότι δέχτηκε τις περισσότερες τροπολογίες μου, ιδιαίτερα για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και την ε, μεταρρύθμιση του συστήματος δικαιοσύνης. Συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να ε, προωθήσουμε το κράτος δικαίου στην Κροατία, να προωθηθεί. Αυτό αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Έχω υποβάλει μια τροπολογία, μια ιδιαίτερη τροπολογία και θα ήθελα να αφαιρθώ περισσότερο σε αυτήν. Στην τροπολογία αυτή υποστηρίζω το μέλημά μας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, προβάλλει συνεργασία με τις κροατικές αρχές έτσι ώστε να υπάρχει ένας εποπτικός μηχανισμός μετά την ένταξη για να δούμε που υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, διαφθορά, απάτη και ούτω καθεξής για να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις να μην αναχαιτιστούν. Αυτός ο μηχανισμός θα ήταν ε, υπέρ του κροατικού λαού, διότι οι Κροάτες θέλουν να συνεχίσουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις και επίσης οι μεταρρυθμίσεις θα ε, ελέγχονται, θα υποπτεύονται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα πρέπει δηλαδή να θεωρηθεί πειθαρχικό μέτρο κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να σας ε, ε, να αναφερθώ στο γιατί δεν είναι τα πάντα έτοιμα η προεργασία δηλαδή. Γνωρίζουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να γίνουν σε ε, ένα τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει εποπτεία και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ως προς σύγκρουση συμφερόντων και έλεγχο, τον έλεγχο ε, τη σύγκρουση συμφερόντων, ξέρουμε ότι το πλαίσιο αυτό δεν είναι ακόμα λειτουργικό. Ελπίζουμε να γίνει στο εγγύς μέλλον. Τα μέλη αυτού του φορέα διορίστηκαν 10 μέρες πριν και γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε αυτό το μηχανισμό. Επίσης, οι πολιτικοί διορισμοί στα Υπουργεία θα πρέπει να προχωρήσουν ε, παραπέρα. Δηλαδή, είναι πολιτικού χαρακτήρα οι διορισμοί περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Οι εποπτικές αρχές ε, σε επιχειρήσεις έχουν αντικατασταθεί με άμεσους διορισμούς. Νομίζω ότι η πολιτικοποίηση δεν ε, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και χρήζει παρακολούθησης. Η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων στη συνέχεια. Οι τροπολογίες δεν είχαν εγκριθεί μέχρι δέκα μέρες πριν και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξει εφαρμογή αυτού του πλαισίου μέσα στα πλαίσια του κοινοτικού ευρωπαϊκού νόμου χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Επίσης δεν ξέρουμε ποια είναι η εποπτική αρχή, ποιος είναι ο βασικός επιβλέπων καταπολέμησης της διαφθοράς και της απάτης ε, αυτό τους τελευταίους έξι μήνες. Όλα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το μηχανισμό. Δεν θέλω να συγκρίνω την Κροατία με τη Ρουμανία, αλλά νομίζω ότι και οι κροατικές αρχές θα πρέπει να βρουν μία διαδικασία παρακολούθησης και οι κροατικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους ε, να μην επεκτείνονται πολύ στις παρεμβάσεις τους. Η κυρία Τάνια Φαγιών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι η Κροατία θα είναι το επόμενο επιτυχημένο παράδειγμα χώρας που προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές ε, ότι για μας η ένταξη της Κροατίας είναι πολύ σημαντική και για τις διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και για τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις. Και είναι πολύ σημαντικό για όλες τις χώρες ε, των Δυτικών Βαλκανίων που χτυπάν την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το μήνυμα ότι η διεύρυνση συνεχίζεται και είναι πραγματικότητα. Φυσικά αυτό εξαρτάται και από τη δέσμευση των ε, κυβερνήσεων. Όπως είπε και ο κύριος Ρότσεκ, η Κροατία έχει σχεδόν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις και ελπίζω ότι η αξιολόγηση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα είναι θετική. Ο πρόεδρος Σλοβενίας, ο Γιάννης Γιάνσα, είχε κάποιες προσδόκητες ε, αντιδράσει ό,τι αφορά τη Λιουμπλιανσκα Μπάνκα. Ελπίζω όμως ε, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην ε, διευθέτηση του προβλήματος και ευελπιστώ ότι στις 11 Μαρτίου στην ε, συνάντηση υψηλού επίπεδου μεταξύ των Πρωθυπουργών θα τεθούν τα θεμέλια για την διευθέτηση αυτής της διαφοράς που δεν είναι μόνο διμερής διαφορά αλλά είναι απόρρια της, των νομικών συνεπειών της διάλυσης της Ιουκοσλαβίας. Δεν ξέρουμε ακόμη ποια θα είναι η κατάσταση στην κυβέρνηση της Σλοβενίας. Πάντως προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι η κύρωση της ενταξιακής συνθήκης και αυτή είναι η επιθυμία και της δικής μου πολιτικής ομάδας. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι πρώτα η Σλοβενική κυβέρνηση και η Σλοβενική Βουλή θα κυρώσουν τη συνθήκη και ότι δεν θα είμαστε η τελευταία χώρα που θα το κάνει. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ρόουτσεκ για την καταπληκτική του προσπάθεια και το πολύ αξιόλογο ψήφισμα. Φυσικά και εμείς ε, συμμετείχαμε ενεργά στις ε, εργασίες για την ένταξη της Κροατίας στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη σταθεροποίηση και την περαιτέρω διεύρυνση. Θα πρέπει η Κροατία να δώσει το παράδειγμα και να μοιραστεί την εμπειρία της με τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Φυσικά πρόκειται για μια διαδικασία που έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα, αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί. Θα μπορούσαμε λοιπόν να απευθύνουμε έκκληση προς κροατικές αρχές να επιμείνουν ιδιαίτερα στην ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που μερικές φορές απειλείται όχι μόνο εκεί, αλλά και σε άλλες χώρες της περιοχής. Ο κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω εγκάρδια και θερμότατα τους συναδέλφους από την Κροατική Βουλή. Συμμετέχουν στη συνεδρίασή μας και γίνονται μάρτυρες των εργασιών της Επιτροπής μας και ευελπιστώ ότι θα είναι αυτή η τελευταία συζήτηση που γίνεται στην Επιτροπή μας για την ε, Κροατία. Εγώ πάντως είμαι πολύ ικανοποιημένο γιατί η Πρωθυπουργοί και της Σλοβενίας και της Κροατίας φαίνεται ότι επιθυμούν να επιλύσουν το κρεμές πρόβλημα της Λιμπλιανσκα Μπάνκα υπάρχουν θετικέ προοπτικές για τη διευθέτηση αυτή τη διαφορά. Εγώ κατέθεσα μια τροπολογία που αφορά αυτή την τελική φάση, την τελική ευθεία τη κροατία ε, ε, στον δρόμο της ένταξης και ελπίζω να ε, εγκριθεί η τροπολογία μου. Μάλιστα κατέθεσα αυτή την τροπολογία για να ενισχύσω αυτό το θετικό κλίμα που επικρατεί στην τελική φάση πριν από την ένταξη και πριν την ε, ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης της ενταξιακής συνθήκης. Όπως είπε και η κυρία Φαγιόν, θα ήθελα να πω ότι εγώ κατανοώ την αντίδραση του Πρωθυπουργού της Σλοβενίας. Θέλει να δοθεί μια αξιόπιστη λύση σε αυτό το εκρεμές πρόβλημα. Και είναι αλήθεια ότι το κόμμα στο οποίο ανήκε ο, ο Υπουργό Εξωτερικών έμεινε εκτός, ε, κυβέρνηση, εκτός κοινοβουλίου. Γι' αυτό έγινε και η αλλαγή του χαρτοφυλακίου που ήταν κάπως ε, απροσδόκητη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον κύριο Ρότσεκ για το υψηλής ποιότητας έγγραφο που συνέταξε που είναι έμπνευση για πολλούς ευρωβουλευτές για να καταθέσουν τροπολογίες. Επιτρέψτε μου πρώτα να τονίσω ότι η Κροατία σημειώνει τον δεκάλογο που περιλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Monitoring Report και τις συγκεκριμένες προσδοκίες που περιγράφονται και στο έγγραφο, άλλωστε, και σας διαβεβαιώ ότι εμείς, οι Κροάτες κοινοβουλευτικοί, που συμμετέσχαμε σε συνεδρίαση με την Υπουργό Εξωτερικών και συμφωνώ μαζί της ότι, ότι τα πράγματα πάνε καλά. και ότι κινούνται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με την ευκαιρία τονίζω ότι οι στόχοι αυτοί δείχνουν και την πρόοδο που έχει επιτύχει η Κροατία στην επίτευξη αυτών των benchmark που ανέλαβε ήδη από την αρχή δηλαδή της διαπραγματευτικής διαδικασίας να εκπληρώσει και ότι αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται. Το νέο αυτό μοντέλο, γιατί πρόκειται για νέο μοντέλο, βασισμένο στις εμπειρίες παρελθουσών εντάξεων με βασική ιδέα ότι η υποψήφια χώρα αναλαμβάνει δεσμεύσεις να είναι πανέτοιμη να αναλάβει όλα τα καθήκοντα από την αρχή της ένταξης. Αυτό έχει γίνει στην Κροατία, αλλά αυτό αποκλείει και το post-taxation monitoring. Επομένως να ζητείτε monitoring για μετά την ένταξη είναι σαν να αμφισβητεί κανείς την επιτυχία του μοντέλου αυτού. Ιδίω με την έννοια ότι η Κομισιόν παρακολουθεί τη διαδικασία αυτή στενά από την αρχή και θα συνεχίσει να το πράττει μέχρι 1η Ιουλίου φέτος η Κροατία. Είναι πολύ σοβαρή ό,τι αφορά τον αγώνα κατά της διαφθοράς. Έχει όντως μεταρρυθμίσει τη δικαιοσύνη της για να ευθυγραμμιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως έχει γίνει και με προηγούμενες ε, εντάξεις. Το κεφάλαιο 23 ήταν το πιο δύσκολο γιατί περιλαμβάνει τις πιο σοβαρές και δύσκολες δεσμεύσεις. Ο κύριος Φιούλε, επίτροπος στις τελευταίες παρατηρήσεις που έκανε, είπε ότι δεν υπάρχουν άλλα εκκρεμή θέματα σε αυτό το κεφάλαιο. Και σε ό,τι αφορά την Λουμπλιάνσκα Μπάνκα, να μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένα εναλλακτικό σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή για την Κροατία. Η Κροατία στην Ένωση, αυτό σημαίνει ότι είναι προς συμφέρον όλων των μερών. Είναι διμερό θέμα η ε, Λουμπιάνσκα μπάνκα και τέτοια διμερή θέματα δεν πρέπει να επηρεάζουν με κανένα τρόπο την πορεία της εντάξεως. Υπάρχει ανοιχτή γραμμή, διάλογος και φαίνεται να διαγράφεται κάποια λύση. Γνωρίζουμε ότι οι όλοι διαδικασία των διαπραγματεύσεων και συζητήσεις όπως η σημερινή παρακολουθούνται από τους άλλους γείτονές μας των Δυτικών Βαλκανίων. Γνωρίζουμε επίσης ότι η διαπραγματευτική μας διαδικασία αποτελεί και πρότυπο για τις άλλες αυτές χώρες. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουν οι χώρες αυτές και μια γενική εικόνα επικοδομητικής συνεργασίας την οποία επιδιώκει η Κροατία και επομένως σαν ένα καλός να ορίσετε ας πούμε προς όλες τις χώρες οι οποίες ενδεχομένως κάποτε θα θέλουν να ενταχθούν. Και στην τελευταία συζήτηση και στη σημερινή οι συνάδελφοί μου ακούω ότι ζητούν από τις χώρες μέλη να κυρώσουν την ένταξη της Κροατίας το δυνατόν συντομότερο. Το παρόν κοινοβούλιο πάντοτε στήριξε την κροατική προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Παρακαλώ, μην λησμονείτε το ρολόι. Το βλέπετε στην οθόνη. Ο κύριος Κράισλερ Ντέρφλερ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος και εγώ, όπως άλλωστε είμαι συνήθως. Βλέπω ότι φοράτε και τα ακουστικά σας πολύ ωραία. Χαίρομαι που σύντομα η Κροατία θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένω πραγματικά πολλά από την ένταξη αυτή. Γνωρίζω την Κροατία και από τις διακοπές αλλά και έχω και πολλούς Κροάτες φίλους. Ακούω να μιλούν για διαφθορά, πολλοί και πολλές. Για μένα το κρίσιμο είναι να λειτουργούν οι θεσμοί, να υπάρχουν οι νόμοι, να λειτουργεί η διάκριση των εξουσιών. Ακούστηκε και για μια τράπεζα, τη Λουμπιάνσκα. Υπάρχει όμως και η Hypo που και αυτή μας διασκεδάζει πολύ εμάς εκεί στη Βαυαρία και άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια θέματα, άκουσα ότι είναι διμερεί Εμεί, στα νυν κράτη-μέλη της Ένωσης έχουμε αρκετά ασχοληθεί με διαφθορά. Ελπίζω λοιπόν η Κροατία να μην μιμηθεί το υπόδειγμα, α πω έτσι, μερικών ήδη χωρών μελών. Α το πω και αυτό λοιπόν. Με χαρά λοιπόν περιμένω την ένταξη της Κροατίας για να μπορέσω να συνεργαστώ και στενότερα και να συζητήσω και με τους συναδέλφους που θα προσέλθουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ράντος.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 Mm-hmm. Mm-hmm. Συνεχίζει ο κύριος Ράντος στα αγγλικά. Θα τονίσω μερικά σημαντικά νομίζω θέματα για την κροατική ένταξη. Η Κροατία μέσα στην, ένταξη, μέσα στην προσπάθεια αυτή έχει ενισχύσει τους θεσμούς της για να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο δημοκρατικών προτύπων και νομίζω ότι επέτυχε η Κροατία στην προσπάθεια αυτή. Και αυτό είναι επιτυχία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα. Η Κροατία θα συνεχίσει να πράττει τα δέοντα και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται ε, στο ψήφισμα, όλα τα θέματα όπως ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο αγώνας κατά της διαφθοράς, η ελευθεροτυπία, θα είναι και δικά μας θέματα. Ταυτόχρονα όμως είναι και η οικονομική σταθεροποίηση, η δημοσιονομική και νομισματική σταθερότητα, καθώς και η δημιουργία των απαραίτητων όρων για τις επενδύσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρότσεκ για το ψήφισμα που συνέταξε και ιδίως για τις συμβαστικές τροπολογίες που βρίσκω πολύ θετικές και που βελτιώνουν το ψήφισμα. Ε, νομίζω ότι αποτελεί επιτυχία του κυρίου Ρότσεκ, αλλά βέβαια και όλων των πολιτικών ομάδων που κατέληξαν σε συμφωνία για την συμβαστική τροπολογία. Ωστόσο δεν μπορώ να υποστηρίξω ορισμένε τροπολογίε που κατά τη γνώμη μου δεν εντάσσονται στο ψήφισμα, όπως για παράδειγμα η θέση και η συμπεριφορά της Καθολικής Εκκλησίας. Συμφωνώ λίγο πολύ με τον κύριο Βάγκελ, νομίζω ότι δεν εντάσσεται στο παρόν ψήφισμα το θέμα αυτό. Υπάρχουν και ορισμένες άλλες προτάσεις νομίζω που είναι κατάλληλε για το ψήφισμα αυτό. Θα ήθελα να πούμε δηλαδή λίγα για την πρόταση η Κροατία να εφίσταται το monitoring και μετά την ένταξη. Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν είναι σωστό, διότι η Κροατία πέρασε μια πολύ απαιτητική διαδικασία διαπραγματεύσεων, πολύ αυστηρή παρακολούθηση, monitoring δηλαδή, στην πρώην ταξιακή περίοδο. Θεωρώ λοιπόν ότι τέτοιου είδου παρακολούθηση δεν θα είναι, δεν θα είναι ορθή για την Κροατία. Η κυρία Ντόρις Πακ. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια και Ρότσεκ πρώτα. Νομίζω ότι αυτό που θα πω τώρα είναι και το κίνητο της κυρίας Μάκοβεϊ. Δηλαδή, διαπιστώσαμε ότι έχουν εφαρμοστεί άλλα κριτήρια στην περίπτωση της Κροατίας. Δηλαδή, χρειάστηκε να περάσει πολύ περισσότερα από τη Ρουμανία και η Βουλγαρία. Και γι' αυτό η Κροατία βρίσκεται σήμερα εκεί που βρίσκεται. Εγώ θεωρώ ότι ναι, μεν εμεί στο κοινοβούλιο τα είδαμε τα πράγματα αυτά, αλλά οι κυβερνήσει δεν τα είχαν δει. Εμείς λοιπόν διδαχτήκαμε ορισμένα πράγματα. Είπαμε ότι οι χώρες μπορούν να ενταχθούν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Και η χώρα σας πληρεί τις προϋποθέσεις. Και πέρσι υποστηρίξαμε την ένταξη της κουρατίας στην Ένωση με το μεγαλύτερο από ποτέ αριθμό βουλευτών. Και τώρα το μοντέλο αυτό που είπατε των διαπραγματεύσεων και στη δική μου χώρα αλλά και στην χώρα του Κράσιλ δεν έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Το monitoring process διαπιστώνει από τα εναπομένοντα 40 είναι ίσως 10 αυτά που μένουν τα οποία θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι Μάρτιο ή Απρίλιο. Και νομίζω ότι το monitoring είναι θετικό για να γίνει δηλαδή μέχρι την ένταξη δεν θεωρώ όμω ότι μια χώρα η οποία θα έχει ενταχθεί πρέπει να γίνεται αντικείμενο διαφορετική μεταχείρισης από άλλε. Τώρα, η διαφθορά βέβαια είναι μέγα πρόβλημα σε όλα τα Βαλκάνια και βέβαια και στην Κροατία. Όχι όμω ότι δήθεν στι άλλε χώρε, τι γειτονικέ σα εκεί, οι οποίε είναι ήδη μέλη τη Ένωση είναι και πολύ καλύτερα τα πράγματα. Άκουσα σήμερα πολλά και για τη Σλοβενία, η οποία υποστήριξε την ένταξη της Κροατίας και άνοιξε η καρδιά μου που το άκουσα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ οι Σλοβαίνοι και οι Κροάτες να διαπράξουν ποτέ το σφάλμα αυτό ενώπιον της ιστορίας, να τηρήσουν δηλαδή μια τέτοια στάση που να μην του επιτρέψει στους μένεις τους δε, να ενταχθούν. Ελπίζω λοιπόν ότι και το θέμα της Λουμπιάνσκα Μπάνκα θα μπορέσει να επιληθεί μέσα και στις υπόλοιπες τις ε, εναπομένουσες διαπραγματεύσεις για το υπόλοιπο της Ιουγκοσλαβίας και ε, να σας πω και το εξή. Η Κροατία δεν θα βάλει και αυτή κανένα εμπόδιο σε καμία άλλη χώρα των Βαλκανίων εφόσον αυτή επιθυμεί να πορευτεί προς μια ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ελπίζω και το αναμένω αυτό και ελπίζω ότι όλοι θα είμαστε και θα φανούμε λογικοί όταν θα θελήσει να ενταχθεί και η επόμενη χώρα. Θα παρακολουθώ πάρα πολύ προσεκτικά το τι θα πράξετε τότε. Χαίρομαι λοιπόν που θα σας δούμε. Thank you, Ms. Park. Now, Ms. Verbat. Verbat. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι λακωνική, γιατί μέχρι στιγμής ε, παρατάθηκε πολύ η συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Ρόουτσεκ, γιατί στην, ε, στο ψήφισμα για την έκθεση παρακολούθηση υιοθετεί μια πολύ θετική στάση για την Κροατία και ευχαριστώ και του και εισηγητέ που φαίνεται ότι συμμερίζονται την άποψη του εισηγητού. Πολλέ φορέ σήμερα αναφερθήκαμε σε διμερεί ζητήματα. Θα ήθελα να τονίσω όπως είπε και η συνάδελφος Doris Πακ, ότι το Κοινοβουλίο ομόφωνα υπερψήφισε μία δήλωση, μία διακήρυξη, που λέει ότι δεν πρόκειται να θέσουμε φραγμούς στις φιλοδοξίες και τα βήματα των συναδέλφων μας από την περιοχή και δεν θα εμποδίσουμε τις ενταξιακές τους βλέψεις, γιατί βιώσαμε πολλές αρνητικές εμπειρίες από την άποψη αυτή. Γι' αυτό και είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να βοηθήσουμε τους γειτονές μας να πραγματοποιήσουν τις ενταξιακές τους φιλοδοξίες. Γιατί είναι αυτό προς το συμφέρον μας, πρώτα απ' όλα, προς το συμφέρον της κρατίας. Σε ό,τι αφορά τη Λιμπλιάσκα Μπάνκα, είναι επίμαχο το θέμα και αφιλεγόμενο όπως ανακούσαμε και σήμερα. Πάντως ε, είμαστε αισιόδοξοι ε, και ευελπιστούμε ότι όταν θα φτάσει το θέμα σε υψηλότερο κλιμάκιο, σε επίπεδο πρωθυπουργών, θα διαθετηθεί εμπρόθεσμα. Συνεχίζονται οι πολύ λεπτέ αυτέ διαπραγματεύσει. Πάντω, ε, ευελπιστούμε ότι θα βρεθεί μία λύση που θα είναι επωφελή και για τι δύο χώρε. Και ελπίζω ότι όλοι θα ικανοποιηθούν με την λύση που θα βρεθεί. Που επαναλαμβάνω, ελπίζω να ληφθεί η συμφωνία αυτή και σε το χρόνο. Σε ό,τι αφορά το μετεξιδα... με... τη μεταξιακή παρακολούθηση, το post-monitoring, Πιστεύω ότι αν εγκριθεί μια τέτοια μετενταξιακή παρακολούθηση θα καταπέσει όλο, όλη η προσπάθειά μας. Γιατί νομίζω ότι υπήρχε ομόφωνη ε, θέση και της Κροατικής Βουλής και μάλιστα υπερκομματική διακομματική συμφωνία υπέρ της ε, ενταξιακής διαδικασίας και υπέρ της ένταξης Κροατίας. Γνωρίζαμε ότι ήταν μακρύς ο δρόμος της ένταξης. Και πραγματικά υιοθετήσαμε με μεταρρυθμίσεις, μεταμορφώσαμε τη χώρα μας, δημιουργήσαμε νέους θεσμούς και σίγουρα δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε τώρα αντίστροφη πορεία. Μην φοβάστε λοιπόν, δεν υπάρχει καμία απολύτω ανησυχία ότι θα αντιστραφεί αυτή η διαδικασία που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ, κύριε Μωρίνοβιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει κυρία Μαρίνοβιτς. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, και κυρίως τον κύριο Ρόουτσεκ. Έχει, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση ε, για την ένταξη της Κροατίας. Είμαστε στην τελική ευθεία, στην πιο αποφασιστική στιγμή και ήρθε η στιγμή να σε ευχαριστήσουμε και να εκφράσουμε τη μεγάλη μας ε, ευτυχία για το ότι θα γίνουμε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε και η συνάδελφος, έχουμε πλήρη επίγνωση της ανάγκης υλοποίησης των υποχρεώσεών μας, της πάταξης της διαφθοράς και της δωροδοκίας, ε, της ε, ενίσχυσης του κράτους δικαίου, αλλά αυτή η διαδικασία είναι ατέρμονη διαδικασία και είναι μια μόνιμη υποχρέωση της χώρας μας. Όπως είπα όμως πριν από λίγο και η Τάνια, η Κροατία είναι πανέτοιμη. Οι πολίτες Κροατίας, ο κροατικός λαός είναι πανέτοιμος να επιλύσει τα προβλήματά του, να διαθετήσει τις εκκρεμότητες με τους ε, γείτονες, ε, με τις γειτονικές χώρες και μάλιστα με ειρηνικό τρόπο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι που δεν το άκουσα ακόμη σήμερα, αλλά καλό θα ήταν να υποθεί. Όπως είπα, έχουμε επίγνωση της να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, τη δωροδοκία, να ενισχύσουμε την απονομή της δικαιοσύνης, να μεταρρυθμίσουμε τη δικαστική εξουσία, να ενισχύσουμε το κράτος δικαίου. Έχουμε επίγνωση όλων αυτών των καθηκόντων μας. Και επίσης θέλουμε πρώτα απ' όλα να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας απέναντι στους συμπολίτε μας, δηλαδή να διαθετήσουμε, να διαφυλάξουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω το το κράτος πρόνοιάς μας. Νομίζω ότι αυτό είναι υποχρέωση όχι μόνο της Κροατίας, αλλά και της ευρύτερη περιοχής. Πιστεύω ότι θα πρέπει ο κόσμος να μας δείξει εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ρόουτσεκ για σύντομα ελπίζω καταληκτικά σχόλια, να ζητήσω από τον κύριο Λάγκε από την Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσετε το λόγο και μια που αναφέρεται η αυστηρή παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενταξιακή διαδικασία, να σας ενημερώσω για, τις, για τα τελευταία επιτέγματα σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση αυτή. Ε, συνεργαζόμαστε στενά με την Κροατία και την αθαρρύνουμε να υλοποιήσει όλες τις ε, κρεμείς υποχρεώσεις της. Θα ήθελα να σας κάνω μια σύντομη σύντομη ενημέρωση για τα θέματα προτεραιότητας που έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η ιδιωτικοποίηση του ναυπηγείου του Σπλίτ. Και χαίρομαι γιατί έχει υποβληθεί ένα θεωρημένο σχέδιο από την Κροατία για την ιδιωτικοποίηση του ναυπηγείου του Σπλίτ και μάλιστα την Τετάρτη θα συνεδριάσει για να εξετάσει το σχέδιο. Βελπιστούμε ότι μετά την έγκριση Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα οριστικοποιηθεί η διαδικασία υπογραφής αυτής της ιδιωτικοποίησης στα τέλη του μήνα. Ένα άλλο θέμα προτεραιότητας αφορά την σύσταση της Επιτροπής για τη σύγκρουση συμφερόντων για τη διαπλοκή. Στις 25 Ιανουαρίου συστήθηκε σχετική επιτροπή και η πρώτη της συνεδρίαση έγινε στις 11 Φεβρουαρίου. Και από αυτή την άποψη λοιπόν έχει η Κροατία τηρήσει την υποσχέωση της. Ό,τι αφορά την ε, δημιουργία σημείο διέλευσης ε, του διαδρόμου Νόιμ στην Αδριατική, θα ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο και εργασία στις 31 Μαρτίου δεν θα είναι έτοιμο δηλαδή τη στιγμή της δημοσίευσης της τελικής μας έκθεσης, αλλά ε, είναι σχεδόν ε, σε τελικό στάδιο και οι εργασίες αυτές. Ό,τι αφορά το θέμα της μετάφρασης, που είναι επίσης ε, προτεραιότητα, έχουμε διαπιστώσει πολύ σημαντική επιτάχυνση της μετάφρασης του κοινοτικού κεκτημένου. Βέβαια δεν θα έχει ολοκληρωθεί η πλήρης μετάφραση του κοινοτικού κεκτημένου την ημέρα δημοσίευσης της ε, τελικής έκθεσης, αλλά αν συνεχιστεί ο ρυθμός αυτός, θεωρούμε ότι όλο το κοινωτικό κεκτημένο θα ε, μεταφραστεί εμπρόθεσμα πριν την ένταξη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Κροατίας και Βοσνίας, την Παρασκευή έγινε μια συνάντηση υπό την Προεδρία του Επιτρόπου ε, Φίλε με συμμετοχή του Υπουργού, της Υπουργού Εξωτερικών Πούσιτς της Κροατίας και του Υπουργού Εξωτερικού της Βοσνίας Ελεζεγοβίνης με θέμα ε, την επίλυση κάποιων εκκρεμών θεμάτων για τα σύνορα μετά την ένταξη. Δεν αφορά διμερεί θέματα σύνοριακά, αλλά αφορά την υποχρέωση της Κροατίας να εφαρμόσει από την πρώτη μέρα της ένταξης το κοινοτικό κεκτημένο. Κάτι που θα δημιουργήσει ίσως προβλήματα στη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Γι' αυτό και έλαβε χώρα αυτή η πολύ επικοδομητική συνάντηση με τους δύο υπουργούς εξωτερικών Κροατίας και Βοσνίας Ερσεγοβίνης, προκειμένου να βρεθούν τρόποι για να διευκολυνθεί η κατάσταση από την πρώτη μέρα ένταξης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρόουτσεκ για να συνοψίσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εντάχει, μετά από αυτή την ε, μακρά συζήτηση, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους για τα σχόλια, νομοδοτήσεις και ούτω καθεξής. Κανείς δεν αμφισβητεί την ετοιμότητα της Κροατίας για να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιουλίου και υπάρχει ευρεία συνένεση όσον αφορά τους συμβιβασμούς. Θα ήθελα να δούμε την πρώτα συμβασμού 2, διότι γνωρίζουμε και εμείς και οι Κροάτες συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση ότι θα συνεχίσει αυτή η εργασία και μετά την 1η Ιουλίου ως προς το κράτος δικαίου κατά πολέμηση της διαφθοράς και ούτω καθεξής. Άρα ζητούμε από τις κροατικές αρχές να επιταχύνουν την καταπολέμηση της κακοδιαχείρισης διαφθοράς απάτης, γνωρίζοντας ότι θα πρέπει να επιμείνουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς, να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα, τη σύγκρουση συμφερόντων και τη διαφθορά. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να εντάξουμε όλες τις ε, γνωμοδοτήσεις σε αυτές τις προτάσεις συμβιβασμού, αλλά δεν συμφωνώ με την πρόταση της κυρίας ε, Μακοβέη ε, ως προς τον μηχανισμό εποπτείας μετά από την προσχώρηση. Όπως είπαν οι Πόσελτ και άλλοι, αυτή είναι το τέλος της διαδικασίας. Εάν εντάξουμε την Κροατία στο μηχανισμό εποπτείας είναι σαν να αμφισβητούμε τη διαδικασία ένταξης. Δηλαδή την πολύχρονη αυτή διαδικασία της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου για τα πεπραγμένα, για τα τεκτενόμενα στην Κροατία. Θεωρώ ότι η Κροατία είναι έτοιμη, ο μηχανισμός υπάρχει, αλλά όπως και σε άλλες χώρες, στη Ρουμανία, στη δική μου χώρα, στη Τσεχική Δημοκρατία και όχι μόνο στα νέα κράτη-μέλη, αλλά και σε πολλά παλαιά θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην καταπολέμηση της απάτης διαφθοράς και ούτω καθεξής. Το να εντάξουμε την Κροατία σε έναν εποπτικό μηχανισμό θα ήταν ένα μείζον λάθος και άδικο για αυτή τη χώρα κατά το τέλος της ενταξιακής διαδικασίας. Θα ήθελα να ε, αναφερθώ στα σχόλια του κύριου Βάιγκελ για την τροπολογία 28. Κατανοώ την άποψή σας, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε σε έναν φορέα ε, στην Καθολική Εκκλησία εμπροκειμένο. Ζητούμε από τις κρατικές αρχές να επαγρυπνούν για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά πολέμηση κάθε ε, είδους ε, διακρίσεων κατά εθνοτήτων, μειονοτήτων, σεξουαλικού προσανατολισμού και ούτω καθεξής. Δεν θα πρέπει όμως να αναφερθούμε σε έναν φορέα και μόνο. Αυτή είναι η έκκλησή μας και νομίζω ότι και οι κροατικές αρχές ε, το γνωρίζουν πολύ καλά. Η κυρία Μπραντνερ, μιλήσατε για την προφορική τροπολογία υπαριθμών 3. Ε, είναι η σωστή κατά την άποψή μας για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ρόλου. Ως προς την κύρωση, διαδικασία κύρωσης χαίρομαι διότι όλοι συμφωνούμε και οι Σλοβαίνοι συνάδελφοι το τόνισαν ότι η διαδικασία κύρωσης θα πρέπει να επιταχυνθεί και στις τρεις χώρες και όταν συναντηθούν οι Πρωθυπουργοί την 11η Μαρτίου θα φτάσουμε σε συμφωνία, δηλαδή θα έχει λήξει και η διαδικασία κύρωσης και από το Σλοβενικό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η άποψη και των Σλοβένων. Θα πρέπει η Κροατία και η Σλοβενία να έχουν αγαστές σχέσεις. Οι δύο αυτές χώρες αποτελούν θετικό υπόδειγμα για τους Σέρβους, Βοσνίους και Μαυροβουνίους. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Ρούτσεκ και όλους όσους συνεισέφεραν σε αυτή τη συζήτηση. Θα ψηφίσουμε, συνάδελφοι, αύριο το απόγευμα για την έκθεση αυτή και τώρα θα στραφούμε στην πρόταση προόδου της Ιρλανδίας μέσα στα πλαίσια της ενταξιακής διαδικασίας. Όπως γνωρίζετε η Ισλανδία διαπραγματεύεται από το 11 και μετά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαπραγματεύσεις συγκινούνται με ταχύ ρυθμό. Από τα μέσα Ιανουαρίου όμως έχουν επιβραδυνθεί οι διαπραγματεύσεις εξαιτία των επικειμένων εκλογών στην Ισλανδία κατά τα τέλη Απριλίου. Υπ' αυτή την έννοια ο εισηγητής μας, ο κύριος Πρέντα, εξέτασε τις 41 ε, τροπολογίες και συμφώνησε με του, του Σκιώδης για 7 ε, τροπολογίες συμβιβασμού. Σας δίνω το λόγο για να μας σχολιάσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. να περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα έτσι ώστε να καθίσουν όλοι όσοι πρόκειται να καθίσουν. Να επικρατήσει ησυχία όπως και να έχει. Μετά το τέλος της διαδικασίας συζήτησης για την ένταξη της Κροατίας. Όπως ε, είπατε, πρόκειται για την έκθεση που αφορά την ενταξιακή και προενταξιακή διαδικασία ε, εισόδου της Ισλανδίας. Ε, στη, το Δεκέμβριο είχαμε και την ε, προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Έχουμε 41 τροπολογίες για τη βελτίωση της έκθεσης και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν τις τροπολογίες αυτές και τους Κιώδης που συνεργάστηκαν μαζί μου για να φτάσουμε σε μία συνένεση όσον αφορά την Ισλανδία. Έχουμε λοιπόν 7 τροπολογίες συμβιβασμού στη συνέχεια που έχουν ε, γίνει δεκτές από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Συναντηθήκαμε στο Στρασβούργο κατά την τελευταία Ολομέλεια και θα ήθελα να σας πω, να σας μιλήσω για αυτά τα κείμενα συμβιβασμού. Καταρχήν, ως προς την παράγραφο 1 του, της πρότασης ψηφίσματος, δηλαδή τη διαδικασία ε, ένταξης και στην παράγραφο 8 για την επιβράδυνση του ρυθμού διαπραγματεύσεων πριν από τις εκλογές του Απριλίου. Ο τρίτος συμβασμός αναφέρεται στην παράγραφο 9, όπου γίνεται λόγος για την κοινή γνώμη της Ισλανδίας ως προς την ενταξιακή διαδικασία και ε, ενισχύουμε το κέντρο πληροφόρησης του Reykjavik και το γραφείο ε, πληροφοριών η τέταρτη πρόταση συμβιβασμού αναφέρεται στις κινήσεις κεφαλαίων και καλύπτει την παράγραφο 13. Ο πέμπτος συμβιβασμός τροποποιεί την παράγραφο 19 που αναφέρεται στον τομέα της αλληλείας και ο έκτος συμβιβασμός ε, αναφέρεται στον αλλιευτικό τομέα και η έβδομη πρόταση συμβιβασμού καλύπτει τη δική μου, μία δική μου τροπολογία, καθώς και τον Τάνον και Άτκινς σε σχέση με την συνεργασία μας στην Αρκτική. Φτάσαμε σε μία επαναδιατύπωση με τρεις προφορικές, μία, δύο και πέντε, και η προφορική ε, τροπολογία 4 αναφέρεται στο, στις αποφάσεις με βάση το iSave και το δικαστήριο 7 και θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να συνεχίσει η καταβολή ε, επιστροφών προς την Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία με βάση την, ε, τις ατασταλίες που υπήρξαν στο iSave. Δυστυχώς, ε, σε σχέση με τον βακαλάο υπάρχουν μεγάλα προβλήματα ως προς τις ποσοστώσεις και δεν φτάσαμε σε συμφωνία με τις όμορες περιοχές και χώρες. Και έτσι η προφορική τροπολογία υπαριθμών 4 αναφέρεται στη μονομερή ποσόστοση βακαλάου που έχει επιβάλει η Ισλανδία. Θεωρώ ότι όλα τα συμβαλόμενα μέρη θα πρέπει να καταβάλουν μία προσπάθεια για εξέβρεση λύσης για να μην έχουμε υπεραλίευση, δηλαδή πλεονασματική αλίευση αυτού του είδους όπως έγινε τα τελευταία χρόνια θα ψηφίσουμε αύριο και στις 13 Μαρτίου θα συζητηθεί το κείμενο, το οποίο θα ψηφιστεί στις 14 Μαρτίου. Συζητήσαμε προγενέστερα το θέμα της Κροατίας. Όταν η Ισλανδία άρχισε τις διαπραγματεύσεις, ορισμένοι συνάδελφοι από την Κροατία ε, είπαν μήπως η Ισλανδία προσχωρεί νωρίτερα από την ε, Κροατία. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Και τότε τους είχα πει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επισυμβεί και ότι, εν πάση περιπτώσει, η κάθε χώρα προσχωρεί με βάση τα δικά της σχετικά πλεονεκτήματα. Η Κροατία θα προσχωρήσει την 1η Ιουλίου, ενώ με το Reykjavik έχει επιβραδυνθεί ο ρυθμός διαπραγματεύσεων εξαιτίας του προεκλογικού, της προεκλογικής εκστρατείας. Τον Απρίλιο θα διεξαχθούν οι εκλογές στην Ισλανδία, αλλά αρκετά πριν αποφασίστηκε η επιβράδυνση του ρυθμού διαπραγματεύσεων. γιατί κρίθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά μέσα στα πλαίσια της ε, προεκλογικής εκστρατείας. Πρόκειται για ένα γεγονός που δεν μπορούμε παρά να καταγράψουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρέντα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω στις 5.30 θα έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ιρλανδίας στη συνεδρίασή μας. Παρακαλώ λοιπόν, ας είμαστε σύντομοι στις παρατηρήσεις μας. Ο λόγος στην κυρία Σάκε, που θα μιλήσει εκ μέρους της Άλδε των Φιλελευθέρων. Είχαμε συναρπαστική συζήτηση για την Κροατία και αυτό δεν πρόλαβα να μείνει ο συνάδελφος ε, που είναι σκιώδης για το θέμα αυτό. Μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω λοιπόν θεωρεί ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προσκόμματα στη διαδικασία. Θεωρεί ότι παρά ε, την ε, έλλειψη της υποχρέωσης, ε, η Ισλανδία συμφώνησε να καταβάλει τα κονδύλια για την iSave. Ο σκιώδης ηγητής συμφωνεί με την έκθεση και αυτά μου ανέθεσε να σας μεταβιβάσω. Ευχαριστώ. Όντως, ήσασταν σύντομοι. Κύριος Ρότσικ. Και εγώ σύντομος θα είμαι, κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους του Γιώργου Φέρμ που επίσης ακολύεται, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή και ισορροπημένη του έκθεση και για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Επίσης να τον ευχαριστήσω για την επικοδομητική του ε, προσέγγιση και την προθυμία να λάβει υπόψη τι δικέ μα τοπολογίε. Είχαμε αρχικά πρόβλημα με το δεύτερο συμβαστικό συμβιβασμό, γιατί θεωρούσαμε ότι δεν θα πρέπει το κοινοβούλιο να αναμειγνύεται ή να σχολιάζει διχόνοια στην ε, Ισλανδική κυβέρνηση. Πάντως η να σχολιαζει διχονια στην ισλανδικη είναι πια πιο σιωροποιημένη, οπότε μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Το μόνο πρόβλημα που μας απέμεινε είναι η συμβαστική τροπολογία 6, ε, η, η τροπολογία 4 και για το ότι ε, εκφράζει την λύπη της για τη μονομερή δήλωση της Ισλανδίας ό,τι αφορά την αλίευση ε, σκουμπριού. Δεν είναι και πολύ επικοδομητική η θέση, η θέση της Ισλανδίας. Θα το σχολιάσουμε αυτό αύριο. Πέραν τούτου όμως ε, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες δεν έχουν πρόβλημα την έκθεση και προσβλέπουμε στην αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των συντηρητικών μεταρρυθμιστών ο κύριος Ρόμπερτ. Ο Σε Ρόμπερτ Άτκινς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέντα για την πολύ ισορροπημένη έκθεση και τον τρόπο με τον οποίο πρωτοστάτησε στις συμβαστικές τροπολογίες και στον τρόπο με τον οποίο διεξήγαγε με τους και οδησηγητές τις συζητήσεις. Ήταν πολύ διαλλακτικός και πρόθυμος. Δεν είναι επίμαχη έκθεση. Υπάρχουν όμως κάποιες επιφυλάξεις και ανησυχίες σε ό,τι αφορά την αλίευση του σκουμπριού και ιδιαίτερα κάποιες αλλιευτικές πτυχές ε, των συζητήσεων. Ο κύριος Τριαν Στίβεσον, πρώην πρόεδρος Επιτροπής Αλίας, όταν μιλάει για, τον, ε, για το σκουμπρί του ανάβουν τα αίματα και πραγματικά φοβίζει τους συνομιλητές, αλλά νομίζω ότι αναγνωρίστηκε αυτή η θέση πια και ότι υπάρχουν προβλήματα με την Αλία και τη Γεωργία. Θα πρέπει και τα δύο κεφάλαια να συζητηθούν εκτενώς πριν καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Πάντως και εγώ συμφωνώ με τον εισηγητή ότι χαιρόμαστε για την θετική κατάληξη των χρηματοπιστωτικών συζητήσεων σε ό,τι αφορά τις χρηματοπιστωτικές δυσκολίες της Ισλανδίας. Πάντως, μόλις το βράδυ άκουσα ένα πρόγραμμα του BBC ένα ημίωρο πρόγραμμα για το πόσο καλά επέλυσε η Ισλανδία τα διάφορα προβλήματα και πόσο λαμπρό είναι το μέλλον της. Τώρα, αν θα, το, το μέλλον της θα εντάσσεται, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να περιμένουμε τις εκλογές ε, και την περαιτέρω ε, συνέχιση της διαδικασίας. Πάντως με την έκθεση του κυρίου Πρέντα δεν έχουμε πρόβλημα, την υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ. Δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο, οπότε να ξαναζητήσω από τον κύριο Πρέντα να κάνει κάποια καταληκτικά σχόλια αν το θέλει. Απλώς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και ιδιαίτερα τους Σκιώδης. Έχω καταγράψει τις επιφυλάξεις που προέρχονται από τους σοσιαλιστές ε, κυρίως. Θα προσπαθήσουμε να εξεύρουμε μία λύση και αν δεν το καταφέρουμε μέσω συμβαστικών θα, γίνει, θα αποφανθούμε μέσω ψηφοφορίας, τελικής ψηφοφορίας. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα λίγη η συζήτηση. Σας υπενθυμίζω ότι θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή αύριο το απόγευμα, όπως προβλέπετε. Και τώρα θα ασχοληθούμε με την ελευθερία του τύπου και το μέσο ενημέρωση ανά τον κόσμο. Η συγγήτρια είναι η κυρία Μαριέτια Σάκε. Όπως γνωρίζετε, αυτή η έκθεση ε, συντασσόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ευτυχώς όμως άρχισε η διαδικασία σύνταξης και τον Ιούνιο θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Και η προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών λήγει στις 9 Απριλίου. Η εισηγήτρια αναφέρθηκε στην προσέγγιση για μη επικάλυψη των εργασιών από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ε, σε σχέση με ζητήματα ε, ελευθεροτυπίας. Επίσης, ε, διεξήγει αυτή την εργασία με τη συμμετοχή όλων, ζητώντας input και στην ιστοσελίδα της βλέπουμε ότι συρρυκνούνται τα δικαιώματα ε, ελευθερίας έκφρασης στις γειτονικές χώρες και πέραν αυτών. Γι' αυτό το θέμα αυτό είναι επίκαιρο. Δίνω το λόγο στην κυρία Σάκε. Σας ευχαριστώ <clears throat> κύριε Πρόεδρε. Όπως εξηγήσατε, είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων στη βάση ενός εγγράφου συζήτηση. Άρα πρόκειται για ένα σχέδιο όπου έχουν ε, συμβάλει και οι stakeholder και η κοινωνία των πολιτών. Βεβαίω και κάθε ένας που είχε την ε, επιθυμία να συμβάλλει με τι σκέψει του. Επομένως, όχι μόνο έγγραφο συζητήσεω. Αυτό που θέλουμε είναι να πάψουμε να βλέπουμε στον τύπο όλες αυτές τις ε, βάναυσες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων μέχρι που φτάνουν μέχρι και φόνο. Η ελευθεροτυπία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της εξουσίας, την ελευθερία της έκφρασης και την πολυφωνία, την πολυφωνική συζήτηση. Και βέβαια, δεν αντιμετωπίζουν μόνο απειλές οι δημοσιογράφοι, υπάρχουν όμως κενές τάσεις που προκαλούνται από την οικονομική κρίση αλλά και από την ψηφιοποίηση που ε, θίγουν ε, τον έγγραφο τύπο και βέβαια το επάγγελμα των δημοσιογράφων. Πώς θα εξασφαλίσουμε την απαραίτητη ποιότητα και αντικειμενικότητα στο έργο του τύπου. Είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προσπαθούμε τώρα να διαμορφώσουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας, να στηρίξουμε και την ελευθερία του τύπου στον κόσμο. Ορόκληρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιοδήποτε, οποιοδήποτε επίπεδο πολιτικής θα πρέπει να ανακατεύεται στην διατύπωση του περιεχομένου του τύπου, αλλά αντίθετα θα πρέπει να διευκολύνει τη δημιουργία πλατφόρμων που να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτές και ελεύθερες. Ε, το έγγραφο αυτό συζητήσεως έλαβε πολλέ εισρωέ από, πολλούς, από πολλά ενδιαφερόμενα μέρη. Δεν είναι όμω πρόθεσή μου, και ελπίζω να συμφωνήσουν οι αδελφοί μου, απλά να επαναλάβω το τι λέει και κάνει η κοινωνία των πολιτών. Γι' αυτό και απεφάσισα να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένε χώρε, διότι σχεδόν σε κάθε χώρα και μάλιστα και σε έναν αριθμό των δικών μας χωρών μελών, αντιμετωπίζουμε προκλήσεις στο έργο αυτό της προστασίας της ελευθερίας του τύπου. Προχωρώ λοιπόν σε μια πιο πολύ θεματική προσέγγιση και Νομίζω ότι πρέπει να τα προωθήσουμε τα θέματα αυτά μαζί και να ακούσω βέβαια και τις απόψεις των συναδέλφων. Από τη μια μεριά βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντική ε, ενίσχυση της θέσης των ανθρώπων και των ατόμων λόγω της ψηφιοποίησης και της ελευθερίας των τύπου, του τύπου και της έκφρασης των σκέψεων και της συμμετοχής στην, σε ανοιχτή συζήτηση και βεβαίως στην του να απευθύνουν, να προκαλούν αυτούς που ασκούν την εξουσία. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και, ε, ε, και ε, πιέσεις κατά δημοσιογράφων που απειλούν αυτούς οι οποίοι ασκούν την εξουσία. Για το λόγο αυτό οι δημοσιογράφοι και τα μέσα αντιμετωπίζουν τις, τους περιορισμού περιορισμούς από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Σε πολλές, πολλές χώρες υπάρχουν και σημαντικές απειλές και μέσω νομοθεσίας με επιβολή προστήμων ή με συγκέντρωση σε λίγα χέρια των μέσων και μάλιστα και σε χέρια πολιτικών ή άλλων που έχουν και συγκρόμενα συμφέροντα. Και μπορούν μάλιστα να οδηγήσουν και σε απειλές κατά της ελευθερίας και μετά την έκφραση. Μάλιστα υπάρχουν και φόνοι δημοσιογράφων ή φυλακίσεις, αλλά και μαζική ε, λογοκρισία που δεν καταπατεί μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις μελιώδεις ελευθερίες, αλλά και το επιχειρηματικό κλίμα. Γι' αυτό θεωρώ ότι η ελεύθερη ροή των πληροφοριών θα πρέπει να είναι κεντρική προτεραιότητα για μας και βέβαια για την ε, προστασία της ελευθερίας του τύπου. Επίσης, ορισμένες οικονομικές εξέλιξεις, όπως η κρίση, η οικονομική κρίση δηλαδή, αλλά και η ψηφιοποίηση, έχουν ενδεχομένως επιπτώσεις στην ελευθερία του τύπου και των δημοσιογράφων, διότι τελικά τα εμπορικά συμφέροντα και τα συμφέροντα του κοινού δεν συμπίπτουν πάντοτε και ιδίως όταν εξετάζουμε το επιγραμμικό περιβάλλον, το online δηλαδή. Ή, διότι ο κόσμος θεωρεί το διαδίκτυο δημόσιο χώρο έκφρασης. Τονίζω επίσης ορισμένες άλλες απειλές που θέτουν οι κυβερνήσεις προς τους δημοσιογράφους και ορισμένους υποστηριχτές των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αναφέρω και τις νομικές πιέσεις ε, λόγω αντιδρομοκρατικών νόμων, αντι, ε, νόμων κατά εξεγέρσεων και ούτω καθεξής. Από την άλλη πλευρά, οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που διαθέτουν ε, με την διοχέτευση διαφημίσεων σε επιλεγμένα όργανα τύπου και ούτω καθεξής. Εγώ κάνω και ορισμένε προτάσει για το πώ μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τα θέματα τη ελευθερία του τύπου ανά τον κόσμο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι για την ώρα. Παρόλο που θέματα ελευθερία τύπου περιλαμβάνονται σε ορισμένα σχέδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ε, Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, υπάρχει κάποια έλλειψη συνοχή στο όραμα αλλά και στα ορόσημα, στα benchmark τα οποία ε, χρησιμοποιούμε. Χρειάζεται λοιπόν μια πιο, πιο, πιο συνεκτική προσέγγιση στο θέμα αυτό ανά τον κόσμο. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη διαφάνεια καθώς και ε, τα κριτήρια που περιλαμβάνουμε στις διάφορες συμφωνίες μας εμπορικές ή άλλες και προγράμματα. Όταν λοιπόν έχουμε, θα έχουμε ξεκάθαρους στόχους κατά νουν, με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερα την εφαρμογή των πολιτικών μας μέσα στα εφιστάμενα ε, εργαλεία όπως, ε, όπως ε, γεωγραφικά ή άλλα. Και αυτά να είναι προσιτά όχι μόνο για μεγάλες οργανώσεις αλλά και για μικρότερους οργανισμούς. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να περιλάβουμε την ανάπτυξη των μέσων του τύπου και την ελευθερία του τύπου σε όλες τις συμφωνίες, να κάνουμε το λεγόμενο mainstream, αλλά και local capacity building, δηλαδή να ενισχύσουμε φορείς ή άτομα τοπικά σε διάφορες χώρες ώστε να μπορούν να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα. Και αναμένω τώρα βεβαίω με ενδιαφέρον τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιακονσάρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια ε, που έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση της κατάστασης και θα ήταν μια και μιλήσαμε για το επιγραμμικό περιβάλλον, είχαμε και μια δημόσια ακρόαση. Αλλά φαντάζομαι θα έχουμε χρόνο να το κάνουμε στο μέλλον. Ο τίτλος αυτός ε, της ελευθεροτυπίας δηλαδή και της ελευθερίας των μέσο μεσικής ενημέρωσης ε, στον κόσμο ε, ε, είναι πολύ φιλόδοξος και θα ήθελα να αναφέρουμε τις χώρες στις οποίες ε, υπήρξε μια δραστική μείωση της ελευθεροτυπίας. Γιατί είναι πραγματικά λυπηρό να συρρυκνώνεται η ελευθεροτυπία και η ελευθερία έκφραση στο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Αν δούμε πάντως τις παγκόσμιες τάσεις γενικώ, διαπιστώνουμε ότι εφόσον οι πολίτες έχουν την ευκαιρία μέσω των κοινωνικών μέσων, των social media να εκφέρουν τη γνώμη τους, δεν πρέπει ταυτόχρονα να συρρυκνώνεται η ελευθερία των παραδοσιακών μέσων μαζική ενημέρωση, γιατί κανονικά οι τάσει αυτέ θα πρέπει να είναι παράλληλε. αλλά αυτή η αντίστροφη πορεία είναι ανησυχητική, γιατί συμβαίνει στι γειτονικέ μα χώρε, στην Τουρκία, στη Ρωσία, ακόμη και στην Ευρώπη. Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, ε, στη Μεγάλη Βρετανία είχαμε διάφορα σκάνδαλα. Βέβαια η Μεγάλη Βρετανία τα ρύθμισε, αλλά και στη Γαλλία και αλλού έχουν χρησιμοποιηθεί διατάξεις ε, κατά της ε, τρομοκρατίας ως πρόσχημα για την περικοπή της ελευθεροτυπίας ή της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν το θέμα πώς η αντιτρομοκρατική νομοθεσία επηρέασε την ελευθεροτυπία, την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η συγκεκριά μας, η κυρία Σάκερ, θεωρεί ότι είναι απόκειται σε εμά, την κοινωνία των πολιτών, να αναλύσουμε το θέμα της ελευθεροτυπίας και ότι θα ήταν σκόπιμο να αφήσουμε ε, να μην κατονομάζουμε συγκεκριμένες χώρες, να μην στυλιτεύουμε συγκεκριμένες χώρες. Εγώ δεν συμφωνώ δεν μπορούμε να αποσιωπούμε καταστάσεις ή να μην ονοματίζουμε χώρες στις οποίες ε, έχει σημειωθεί σημαντική συρρήκνωση το, της ελευθερίας τύπου. Στην Τουρκία, για παράδειγμα, έχουμε τους περισσότερους φυλακισμένους δημοσιογράφους στον κόσμο. Η κατάσταση είναι τραγική. Έχουμε πολύ καλές τροπολογίες, για παράδειγμα μια κοινή πανευρωπαϊκή στρατηγική, και επίσης να δούμε και το θέμα των διεθνών συμφωνιών και της αιρεσιμότητας που θα μπορούσε να συνοδεύει τις συμφωνίες μας ε, για την ελευθεροτυπία δηλαδή και την ελευθερία λόγου. Γιατί λέμε να εξαρτώνται ε, οι συμφωνίες μας ε, να λαμβάνουν υπόψη και τις ελευθερίες αυτές, αλλά μόνο λέμε και δεν κάνουμε τίποτα. Εγώ είμαι ε, εισηγήτρια για το Καζακστάν και διαπιστώνω ότι το Καζακστάν έχει αποδεχθεί τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά αμέσως μετά η Λέδη Άστον ταξίδεψε στην Κεντρική ε, Ασία, πήγε και στο Καζακστάν. Είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και το αναφέρω. Και ήταν μεγάλη απογοήτευση το γεγονός ότι η Λέδη Άστον δεν αναφέρθηκε στις παραβιάσεις της ελευθεροτυπίας, γιατί το Καζακστάν είναι μια χώρα όπου ε, ουσιαστικά η ελευθεροτυπία είναι ανύπαρκτη. Έχουμε και εντεταλμένο πια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρώ ότι η ελευθεροτυπία είναι από αναφέρετα θεμελιώδη δικαιώματα και θα πρέπει ε, για τα θέματα αυτά να έχουμε μια ενιαία φωνή. Το έγγραφο εργασία νομίζω παρουσιάζει πολύ εύστοχα τα προβλήματα, μας δίνει τροφή για σκέψη, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να προτείνει και πιο συγκεκριμένα μέτρα, πιο απτές προτάσεις ώστε να είναι πιο συνεπής και ο τρόπος αντίδρασης Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τέτοια θέματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριο Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το έγγραφο αυτό εργασία, γιατί αν κατάλαβα καλά, περί αυτού πρόκειται, περί ενό εγγράφου εργασία δηλαδή απλώ, νομίζω ότι αγγίζει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα τη ελευθεροτυπία και τη ελευθερία των μέσων μεσική ενημέρωση, ε, που έχουν ζωτικό ρόλο για οποιοδήποτε δημοκρατικό καθεστώς Αρκεί να εξετάσουμε την έκθεση τη Επιτροπής μας για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο κάθε χρόνο και τη λίστα των βραβευθέντων με το βραβείο Ζαχάροφ. Εξετάζοντα όλα αυτά, διαπιστώνουμε τι τραγικέ παραβιάσει ε, της ελευθερίας του βιώνουν οι δημοσιογράφοι στον κόσμο και όχι μόνο σε χώρε που βρίσκονται σε μεταβατική διαδικασία προ τη δημοκρατία, αλλά και αλλού. Νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και όλα τα θεμελιώδη ζητήματα που δημιουργούνται όχι μόνο για τα κλασικά, τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωση, αλλά και για τα νέα ηλεκτρονικά μέτρα που αναφέρει η συγκέντρια είναι πολύ σημαντικά. Και για τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πολύ περίπλοκα και μάλιστα σε κάποιες χώρες, χώρες της Αραβικής Άνοιξης, κάποια πολιτερχικά καθεστώτα εμποδίζουν την ελευθερία έκφρασης στο διαδίκτυο και άλλες ελευθερίες. Και αν εξάρτητα με την ψηφιακή διάσταση την οποία πραγματεύεται η έκθεση, καλό θα ήταν να δούμε ποια είναι η γνώμη όχι μόνο των χρηστών του διαδικτύου, αλλά και ε, εκπροσώπων των επαγγελματιών ε, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και το σχέδιο της προλαλήσας σας, ε, ίσως το σχόλιο της προλαλήσας σας είναι ίσως ενδιαφέρον. Να δούμε τι γίνεται με χώρες που συστηματικά παραβιάζουν αυτά τα δικαιώματα ελευθερίας έκφρασης ε, και την ελευθεροτυπία και την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και ακόμη και στην ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καλό θα ήταν να κατονομάζονται συγκεκριμένες χώρες που κατάφορα παραβιάζουν τέτοιου είδους ελευθερίας. Επίσης, πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την εισηγήτριά μας να είναι πιο συγκεκριμένη σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα και τις προθεσμίες με βάση τις οποίες θα υποβάλει την έκθεση της στην Επιτροπή. Γιατί το βασικό δεν είναι να γίνει μόνο η ανάλυση της κατάστασης. Πάνω από όλα στόχος της έκθεσης, όπως λέει και στο σχέδιο ε, εργασίας της, είναι ποια θα είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εξασφαλίσει απρόσκοπτη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων ε, στις διάφορες πολιτικές της. Αυτή είναι η μόνη κριτική που θα μπορούσα να κάνω στην έκθεση. Θα πρέπει να είμαστε πιο επιφυλακτικοί, πιο, πιο συνετοί με τα λόγια που χρησιμοποιούμε. Εκεί που λέει η, Ευρωπα... η... η κυρία Συγγέντρια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να διαπαιδαγωγήσει κυβερνήσεις. Καταλαβαίνουμε τι εννοεί, αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε πατερναλιστικοί και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή της, δόκιμη, της πιο δόκιμης διατύπωσης. Επαναλαμβάνω, ε, το έγγραφο εργασίας ε, από ενό σημαντικού θέματος, της ελευθερίας, στην πληροφορία και στις ελευθερία στο μέσο μαζικής ενημέρωσης, είναι, θα είναι μία από τις βασικές εκθέσεις ε, συμβολικές για την κοινοβουλευτική μας αιτία. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ ε, σωστή στην απάντηση που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα τα προγράμματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γιατί όχι να μην ε, ε, εγκρίνουμε και ένα ειδικό πρόγραμμα για την ελευθερία στα πλαίσια των διαφόρων δράσεων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, θα ήθελα να σας πω ότι η δεύτερη εξέταση του σχεδίου έκθεσης θα γίνει στις 20 Μαρτίου η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι η 9η Απριλίου, όπως είπα και στην αρχή. Η εξέταση των τροπολογιών στην Επιτροπή μας θα γίνει στις 6 Μαΐου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας την επόμενη μέρα, την 7η Μαΐου δηλαδή. Κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφιστεί η έκθεση αυτή στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Επίσης ε, θα ψηφιστει η αυτη στην επί ευκαιρία να απευθύνω έκκληση προς τις πολιτικές ομάδες να ορίσουν τους εισηγητές τους ε, για την έκθεση πρωτοβουλίας. Και η κυρία Σχάκη για να ολοκληρώσει. Θα είμαι όντως σύντομη. Νομίζω ωστόσο πρέπει να απαντήσω στα σχόλια των κυρίων Γιακονσάρη και Σαλαφράνκα. Γενικά συμφωνούμε, νομίζω. Αναφέρθηκα και εγώ στην χρήση αντιτρομοκρατικών και άλλων νόμων κατά χρηστικό τρόπο, για περιορισμό δηλαδή της ελευθερίας του τύπου, συμφωνώ και με τα όσα είπαν οι δύο συναδελφοί μου ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ορισμένες χώρες όταν υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Για το έγγραφο συζητήσεως προτίμησα να μην αναφέρω ε, συγκεκριμένες χώρες γιατί αλλιώ θα έχουμε ένα τεράστιο κατάλογο, ατελείωτο. Όμως για, στην, ε, ε, στην ε, επερχόμενη συζήτηση χώρες όπως η Τουρκία που είναι σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την πολιτική μας διεύρυνση γενικότερα, είναι σημαντικό να τα πούμε τα πράγματα αυτά γιατί έχουμε και ιδιαίτερη ευθύνη και ευκαιρία να τα πούμε αυτά εκεί. Το ίδιο ισχύει για όρους, ερεσιμότητα δηλαδή, σε εμπορικές συμφωνίες και άλλα. Θεωρώ και εγώ ότι είναι ουσιώδης η αξιοπιστία της Ένωσης. Πρέπει να μιλήσουμε λοιπόν για αιρεσιμότητα και για ειδική στόχευση όπου απαιτείται. Για τα σχόλια του κ. Σαλαφράνκα τώρα πιο συγκεκριμένα που εν μέρη νομίζω απηχούν και τις δικές μου σκέψεις, δέχομαι τα σχόλιά του για την ευαισθησία ορισμένων γλωσσών ή μάλλον ορισμένων διατυπώσεων, για το ευαίσθητο μάλλον ορισμένων διατυπώσεων και επίσης την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών των ε, ρυθμιστών αλλά βέβαια και για την αντιμετώπιση καταστάσεων σε χώρες ή περιοχές που βρίσκονται σε μεταβατικές περιόδους. Επίσης θα εξετάσω για το εάν μπορεί να γίνει κάποια αξιολόγηση μέσα στις εκθέσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων και αλλού. Βεβαίως θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους και νομίζω μέχρι τις 5 Μαρτίου θα πρέπει να υποβάλλετε τις παρατηρήσεις σας αν θέλετε να τις περιλάβω στο πρώτο σχέδιο. Thank you very Εδώ ολοκληρώνεται η εξέταση αυτού του θέματος της ημερησίας διατάξεως και προχωρούμε τώρα στη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Εδώ πρόκειται για την πρώτη εξέταση του σχεδίου εκθέσεως για τη Βοσνία Ριζεγοβίνη τελευταίο από τα εννέα ψηφίσματα φέτος για ε, διάφορες υποψήφιες χώρες. Η χώρα αυτή κινδυνεύει να υστερήσει κατά πολύ από τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, διότι η πρόοδος στην διαδικασία εντάξεως είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Μέχρι τώρα δεν έχει μπορέσει να, εκπληρώσει, να, να επιτύχει τα ορόσημα, τα benchmark που να απαιτούνται για να προχωρήσει η ενταξιακή ε, διαδικασία και να υποβάλει αξιόπιστη αίτηση για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βασική μας ανησυχία παραμένει η ίδια για πολλά χρόνια, δηλαδή η έλλειψη κοινού οράματος της πολιτικής, της ηγεσία για την συνολική μελλοντική κατεύθυνση που θα λάβει η χώρα. Θα δώσω το λόγο τώρα στην εισηγήτρια κυρία Πακ για να εξηγήσει τα βασικά πορίσματα τη εκθεσής. Ε, λίγο πολύ τα είπατε όσο ήταν να πω. Κύριε Πρόεδρε, τι να σας πω άλλο εγώ. Τέλος πάντων. Όλοι γνωρίζετε ότι την προηγούμενη άνοιξη συντάξαμε την πιο πρόσφατη τελευταία έκθεση δηλαδή. Εγώ περίμενα τότε με τη σύνταξη της έκθεσης μέχρι να μπορώ να πω και κάτι θετικό. Το ίδιο ήθελα και φέτος, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνω βρισκόμαστε ακόμα ή πάλι εκεί όπου νομίζαμε ότι είχαμε καταφέρει να προχωρήσουμε την προηγούμενη άνοιξη. Η χώρα είναι διασπασμένη. Βέβαια είναι και η κληρονομιά του Ντέιτον που εμποδίζει να ενωθεί ένα σύνταγμα που δεν το έφτιαξε η ίδια αλλά κάπου το ε, συναρμολόγησαν στο Ντέιτον και η κληρονομιά αυτή είναι βαριά. Έτσι είναι. Υπάρχει εδώ και χρόνια μια απόφαση του δικαστηρίου του Στρασβούργου η χώρα αυτή να αφαιρέσει τις διακρίσεις από το Σύνταγμά της. Βέβαια, αυτά τα έχει βάλει η διεθνής κοινότητα, δεν τα έχει βάλει η ίδια. Αυτή η απόφαση στην υπόθεση σε τη Φίντσι λέει ότι οι, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν και όποια προέλευση και αν έχουν, ότι μπορούν να καταλάβουν επίσημη ε, δημόσια θέση, ακόμα και την ανώτατη. Και όμως δεν γίνεται. Αν δεν είσαι Βόσνιος ή Σέρβος, τότε είσαι ασάς, δηλαδή δεν είσαι τίποτα. Είσαι σαν να ε, είσαι μηδέν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε μια δημοκρατία που βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης, λίγο πολύ. Γίνεται όμως διότι το σύνταγμα αυτό, το οποίο δεν το φτιάξαν οι ίδιοι οι κάτοικοι της Βοσνίας και της αλλά λίγο πολύ, όπως είπα, συναρμολογήθηκε με μεγάλη ταχύτητα τότε στη συμφωνία που οδήγησε στο τέλος του πολέμου. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση τώρα που οι άνθρωποι καλούνται να λύσουν προβλήματα που δεν προκάλεσαν ίδιοι. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η χώρα είναι χωρισμένη σε δύο μεγάλα τμήματα, σε δύο οντότητε, από τη μια δηλαδή την Ρεπούμπλικα Σρέψκα, όπου κυρίω κατοικούν Σέρβοι, και από την άλλη μεριά η Κροατική Μουσουλμανική Ομοσπονδία, κυρίω Βόσνη λοιπόν και 10-12 100 Κροάτες. Το πρόβλημα αυτής της Ομοσπονδίας είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει διότι είναι δομημένη σύμφωνα με την συμφωνία της Ουάσιγκτον του 1994 με τρόπο που είναι αδύνατο να αναλυφθεί οποιαδήποτε πολιτική δράση. Υπάρχουν οι διάφορες τοποθεσίες και τα διάφορα καντόνια με 10 συνολικά πρωθυπουργούς και ένα σμάρι ολόκληρο υπουργού και άλλους και παραπάνω από αυτούς είναι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και ακόμα παραπάνω είναι η κορυφή του κράτους. Επομένω, όντως και, και μόνο λόγω της δομής αυτής δεν προχωρεί τίποτα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι δυσχερέστατο και το λέω από την αρχή, διότι μέχρι τώρα κανένας δεν προσπάθησε να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς εκεί να αλλάξουν τις δομές αυτές. Τα πράγματα έτσι είναι, από το 1996. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι που ζουν εκεί και είχαν ή κατήχαν ή κατέχουν θέσεις, α, λένε μια χαρά είμαστε. Δεν παρετούμεθα από τη δομή αυτή, διότι πολλοί θα μείνουν χωρίς δουλειά. Πολιτικοί θα μείνουν χωρίς δουλειά, αξιωματούχοι θα μείνουν χωρίς δουλειά, ούτως ή άλλως βέβαια, περί τι είναι. Το πρόβλημα λοιπόν είναι μέγα και εμείς δεν φροντίσαμε. Η Κομισιόν δεν φρόντισε και δυστυχώς μόνη που τα φωνάζει αυτά τα πράγματα εδώ και χρόνια είμαι εγώ και κανένα δεν ή το πολύ πολύ προκαλώ έχθρες. Στο μεταξύ επιλήφθηκε του θέματος ακούει. Ή το πολύ πολύ προκαλώ έχθρες. Στο μεταξύ επιλήφθηκε το θέματος η Αμερικανική κυβέρνηση. Είπε «Α, εμείς θα τα φτιάξουμε». Θα λύσουμε τα προβλήματα αυτά έξωθεν. Δεν είναι δυνατόν ωστόσο σε μια χώρα που έχει περάσει δημοκρατικές εκλογές ξανά και ξανά να τα λύσει απ' έξω. Οι άνθρωποι πρέπει να τα δουν τα προβλήματα μόνοι τους και αν θέλουν να ζητήσουν τη, τη βοήθειά μας. Έχει, έχει καλώς. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το μην τα αφήσετε στους Αμερικάνους. Το Dayton φτιάχτηκε στην Αμερική και δεν λειτουργεί. Ευτυχώς βέβαια οδήγησε στο τέλος του πολέμου, αλλά τίποτα παραπάνω. Το πρόβλημα, το πρόβλημα στην Βοσνία Ζεγοβίνη είναι ότι η χώρα μπαίνει όλο και περισσότερο στο τέλμα των εθνικών διαφορών, δηλαδή τα χάσματα μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών μειονοτήτων βαθαίνουν και οι πολιτικοί τα εκμεταλλεύονται αυτά όλο και περισσότερο και τα εντείνουν διότι όλοι επικαλούνται τις διαφορετικές εθνικές τους ιδιαιτερότητες και κάνουν ό,τι μπορούν. Συχνά δεν κάνουν απολύτως τίποτα, αλλά στον τομέα της διαφθοράς εκεί τα πάνε πολύ καλά. Πρόκειται για μια διοίκηση η οποία δεν είναι ιδιαίτερως λειτουργική Όπως λέχθηκε και πριν υπάρχει μεγάλη διαφθορά και είναι και επόμενο εφόσον υπάρχουν τόσο πολλά διοικητικά επίπεδα σε αυτή την χώρα. Εκεί πρέπει να γίνει κάποιος κοινό αγώνας. Τέλος πάντων, την προηγούμενη άνοιξη και μετά από ένα-ενάμιση χρόνο καταλήξαμε να έχουμε μια κυβέρνηση στη Βοσνία Ρεσεγοβίνη, η οποία στη διάρκεια του καλοκαιριού πάλι κατακαιρματίστηκε, διαλύθηκε. Από τον Οκτώβριο υπάρχει τώρα ένα Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι καν κυβέρνηση στο συνολικό ας πούμε, κρατικό επίπεδο. Στο μεταξύ, ωστόσο, έχει διαλυθεί η κυβέρνηση της Ομοσπονδίας Κροατών και Μουσουλμάνων και δεν προχωρεί τίποτα. Ίσως να μην θυμάστε πλέον ότι η χώρα αυτή δεν μπορεί να κρίνει και να αποφασίζει μόνη της. Εξακολουθεί να έχει, είπα το εκπρόσωπο, που δεν είναι εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς στείλαμε εκεί τέτοιον πέρσι υπάρχει ένα σημαντικός πρέσβης, ο κ. Σόρενσεν, της Λέδης Άστον δηλαδή, που εκπροσωπεί στην χώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι όμως απλά αρχηγός αντιπροσωπείας, έχει άλλο καθεστώς. Το πρόβλημα είναι ότι εκτός από αυτόν υπάρχει και ένας high representative, ο οποίος είναι υπόλογος στη διεθνή κοινότητα, δηλαδή και σε Ρώσους, Αμερικανούς και όλους. Αυτός ο θεσμός που λειτουργεί, υπάρχει τέλο πάντων από τα μέσα της δεκαετίας του 90 για να συνδράμει στην ανοικοδόμηση της χώρας και να εμποδίσει τη δράση πολιτικών οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα συμφέροντα. Αυτός ο ύπατος πρόσωπος εξακολουθεί να διαθέτει, να έχει μάλλον την αρμοδιότητα να φροντίζει για την εφαρμογή της συμφωνίας του Dayton, έχει μάλιστα και νομοθετικές αρμοδιότητες και όντως εκδίδει νομοθετήματα. Εφόσον δεν συμφωνούν οι πολιτικοί, τότε αποφασίζει ο ύπατος πρόσωπος. Τότε οι πολιτικοί βέβαια μπορούν να πούν «Α, εμείς νύπτουμε τα σχήρα μας». Μα έτσι δεν μπορεί να ασκηθεί υπεύθυνη πολιτική και να ανθίσει μια χώρα. Και αυτό ο ύπατος εκπρόσωπος ε, λέγω, εξακολουθεί να υπάρχει και θα μείνει άλλωστε εκεί στο πόστο αυτό μέχρι ότου επιληθούν και τα τελευταία θέματα που προκύπτουν από το Σύνταγμα. Έχουμε λοιπόν μια πραγματικά αξιοθρύνητη κατάσταση, σχεδόν καθόλου επενδύσεις, επίσης για τον λόγο ότι για να γίνουν επενδύσεις πρέπει να είναι ορατό και ένα κράτος δικαίου και μια διοίκηση. Το πρόβλημα είναι όμως ότι στο ένα επίπεδο, ας πούμε σε μια κοινότητα έχει τα ενία ένα κόμμα, αλλά στο καντόνι στο οποίο ανήκει αυτή η κοινότητα έχει τα ενία της εξουσίας στο χέρι άλλο κόμμα και έτσι δεν προχωράει τίποτα. Υπάρχει μια τέτοια κατάσταση για την οποία δεν ευθύνονται όλοι αυτοί βέβαια, αλλά η οποία υπάρχει. Μετά είναι, μπαίνει και το θέμα της εκπαίδευσης, που εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Για να προσελκυστούν επενδύσεις και επενδυτές, χρειάζονται και καλά εκπαιδευμένοι νέοι άνθρωποι. Στη χώρα αυτή ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει μια κατάσταση που λέει δύο σχολεία κατά την ίδια στέγη. Από την αριστερή πλευρά μπαίνουν οι καθολικοί, από τη δεξιά οι μουσουλμάνοι. Αυτά είναι μεσαιωνικές καταστάσεις. Έτσι προκαλείται μονάχα έχθρα. Δεν καταλήγουν στη συμφιλίωση ούτε βέβαια σε ένα ενιαίο κράτος ξεκολουθούν να υπάρχουν αντιθέσεις και γι' αυτό βέβαια δεν έρχονται και αλλοδαποί επενδυτές. Δεν υπάρχουν λοιπόν τα απαραίτητα για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να μπορέσουν έτσι να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανεξάρτητα τώρα και από το θέμα του Κόσοβου είναι και το τελευταίο, ο τελευταίος κρίκος σε αυτή την κοινότητα δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτό μπορώ να το πω. Δεν προχωρούν σε κανένα τομέα. Ορισμένα νομοθετήματα όντως ήδη εκδόθηκαν, όπως ο νόμος για τη λογοκρισία, επίσης οι προϋπολογισμοί. Αλλά το πολιτικό τοπίο είναι τόσο κατακαιρματισμένο και είναι τόσο διαβρωμένο από πολιτικές, προσωπικές έχθρες, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρηθεί αυτή η χώρα ως ενία. Κοιτάξτε, 13 Υπουργοί Παιδείας. Ε, πώς να λειτουργήσει το σύστημα εκπαίδευσης. Στη χώρα υπάρχουν 167 Υπουργοί στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Μα αυτοί τρώνε όλο τον προπολογισμό. Δεν γίνεται και διαφορετικά. Άρα, πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα εάν δεν ρίξουμε το βάρος μας στα συγκεκριμένα, στα πιο σημαντικά πράγματα. Για παράδειγμα, στήριξη τη της αστυνομίας. Εκεί είναι και το ΝΑΤΟ βέβαια, με την Ανθέα, με την αποστολή Ανθέα. Αλλά αυτά είναι βοήθειες. Αλλά δεν είναι η βοήθεια που προσφέρει δυνατότητα αυτοβοήθειας, δηλαδή να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Δεν θα θρυνήσω περισσότερο γιατί νομίζω σε πέντε λεφτά έχουμε εδώ υψηλό προσκεκλημένο, αλλά διαβάστε το κείμενο, δεν είναι και ιδιαίτερα μακροσκελές, μπορούμε να το κάνουμε και πιο έντονο αν θέλετε. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως είναι αρκετά έντονο. Το άσχημο είναι ότι σήμερα ε, λέγω τα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είχα πει και ήδη πριν από ένα χρόνο. Δηλαδή δεν βλέπω πρόοδο. Και αυτό είναι το λυπηρό, διότι αυτοί που υφίστανται όλα αυτά είναι οι νέοι. Κυρίως αυτοί που θίγονται από αυτά είναι οι νέοι οι οποίοι εν τέλει ζητούν καλύτερη τύχη στην αλλοδαπή. Και έτσι αυτό το περίφημο brain drain, το άδειασμα των εγκεφάλων, είναι σημαντικό. Είναι πάρα πολύ έντονο στη χώρα αυτή. Αυτό, αυτή την τάση θα έπρεπε να κάνουμε προσπάθεια να την αντιστρέψουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν ακόμα μεγαλύτερη δέσμευση, ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και του δικού μας εκπροσώπου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. Νομίζω τα γνωρίζει αυτά και η Κομισιόν και ελπίζω πολύ ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή και σε ένα σημείο ώστε και ο ύπατος εκπρόσωπος της διεθνούς κοινότητας να μπει στο αρχείο πλέον και να μπορέσουν οι άνθρωποι εκεί να σταθούν στα πόδια τους. Αυτό είναι επίσης αίσθημα ευθύνης. Κύριος ε, θα ήθελα να πω ότι η έκθεση είναι εξαιρετική, αλλά δυστυχώς ε, είναι λυπηρό αυτό το ανάγνωσμα, διότι υπάρχει έλλειψη προόδου, θα θέλαμε περισσότερη, αλλά υπάρχουν ορισμένοι προγενέστεροι όροι, ορισμένες προϋποθέσεις για να δούμε πώς θα λειτουργήσουν οι θεσμοί θα πρέπει να υπάρχει συνένεση ε, ως προς την ενταξιακή διαδικασία. Επειδή υπάρχουν ε, λοιπόν αυτές οι διαφορές και οι διχασμοί, είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα. Θα υποβληθούν και τροπολογίες στη συνέχεια όσο αφορά το οικονομικό σκέλος, υπάρχει μία συμφωνία για την προσχώρηση της ε, Βοσνίας των ε, ΠΟΕ, άρα υπάρχουν ε, ενθαρρυντικά στοιχεία στην έκθεση αυτή. Το ίδιο ισχύει όταν μιλάμε για την παράγραφο 27. Ακούσαμε ότι έγινε αυτή η συνάντηση μεταξύ Επιτρόπου Φίλε και των Υπουργών Εξωτερικών από τις δύο πλευρές. Αυτά είναι θετικά παραδείγματα τα οποία μπορούν να ενταχθούν στην έκθεση για να ενθαρρύνουμε τους Βόσνιους φίλους να εργαστούν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ελπίζουμε να συμβεί κάποια στιγμή, να γίνει κάποια στιγμή. Η κυρία Λούνατσεκ εντάχει. Ε, αντικαθιστώ τον, την κυρία Κορνέλισεν και όπως είπε και ο κύριος Ρούτσεκ και η, η έκθεση αυτή είναι πολύ καλή, όχι αισιόδοξη βεβαίως. Είπατε ότι η συμφωνία ε, Dayton σταμάτησε τον πόλεμο αλλά δεν έφερε την ειρήνη μακροχρόνια. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα στα οποία θα ήθελα να σταθώ εντάχει ως προς την οικονομική κατάσταση. Καταρχήν, αναφερθήκατε στα προβλήματα των νέων, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι η ολόκληρη περιοχή έχει ε, πληγεί και από την κρίση, τη δική μας κρίση, ιδιαίτερα στη Βοσνία, διότι το νόμισμά τους συνδέεται με τον ευρώ και δεν μπορούν να το υποτιμήσουν. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό με μία τροπολογία. Ως προς την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους Βόσνιους να έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Ιδιαίτερα δύσκολο και πιο δύσκολο από κατοίκους ε, τρίτων χωρών που δεν βρίσκονται στη διαδικασία διεύρυνσης. Μιλήσατε και για την κατάσταση των γυναικών, ε, την ε, βία στο σπίτι. Αυτό το θέμα θα πρέπει να μας απασχολήσει όχι μόνο στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, αλλά και σε, άλλα, και σε άλλες περιφέρειες των Βαλκανίων. Στο 9 μιλάτε για την απλούστευση της ε, διάρθρωσης ε, της ε, Βοσνίας Ερζεγοβίνης σε καθαρά εθνοτικό επίπεδο και θεσμικό, αλλά δεν είναι, πάρα πολύ, δεν είναι εύκολο αυτό για τη Βοσνία Αρζεγοβίνη. Ως προς το 25 για, για, το σύστημα ασύλου, ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δικαίωμα ε, πρόσβασης και ταξιδιού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το καθεστώς free travel, θα ήθελα να υποβληθεί μια τροπολογία έτσι ώστε να ζητηθεί από τα κράτη-μέλη να προβλέψουν διαδικασίες για τους ετούντες άσυλο, έτσι ώστε οι διαδικασίες να είναι πιο γρήγορες από ό,τι μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ και πιστεύω εξ ονόματος της κυρίας Κορνέλισεν ότι θα υπάρξει αγαστή συνεργασία με τους ε, σκιώδεις. Σας ευχαριστώ. Και ένα λεπτό για την κυρία Παμπαλώνη, που είναι Ματάρχης της Γενικής Διεύθυνσης ε, Διεύρυνσης. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την κυρία Πακ για την πολύ καλή της, πολύ εύστοχη έκθεση. Η Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως ε, την ανάλυση που κάνει στην έκθεσή της η κυρία Πακ, γιατί Τη συνάδει με τη δική μας αξιολόγηση στην ετήσια έκθεση πρόοδου του Οκτωβρίου για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Δυστυχώς ε, δεν ήταν πολύ θετικό το συμπέρασμα και της δικής μας αξιολόγησης. Είναι αρνητικέ εξελίξεις. Μια και έχουμε ελάχιστο χρόνο, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρία βασικά σημεία του διαλόγου που έχουμε με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη που αναφέρονται και στην έκθεση της κυρίας Πακ. Ε, έχουμε την, ε, το διάλογο υψηλού επίπεδου για την προταξιακή διαδικασία με δύο πρωταρχικούς στόχους, ε, την αρρωγή για την, στη δικαστική εξουσία προκειμένου να εφαρμοστεί η νομολογία σε και έχουμε πολύ έντονο διάλογο και με τους πολιτικούς ηγέτες προκειμένου να ε, διευκολύνουμε την ανέβρεση λύσης ε, μεταξύ των πολιτικών αρχηγών προκειμένου να υποβληθεί μία πρόταση στην ε, Βοσνιακή Βουλή για να περάσουμε στο δεύτερο επίπεδο και να εφαρμοστεί πλήρως η Συμφωνία Σύνδεσης και Σταθεροποίησης που είναι προϋπόθεση μιας αξιόπιστης υποψηφιότητας της Βοσνίας για ένταξη που θα λάβει χώρα μετά την συνταγματική αναθεώρηση. Και μάλιστα στο γραφείο μας στο Σαράγεβο ε, στείλαμε επιστολή ε, της Λέδη ε, Άστον και του Επιτρόπου Φίλε προς όλους τους πολιτικούς αρχηγούς προκειμένου να επιτεχηθεί κατεπηγόντως η εφαρμογή της σχετικής δικαστικής απόφασης. Επίσης έχουμε δεύτερο διάλογο υψηλού επίπεδου για την ε, δικαιοσύνη. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει τον Απρίλιο στην επαρχία Βέρσκομ είναι πολύ σημαντικό με τις προσπάθειες ε, που κάνουμε στη Βοσνία Ερζεγοβίνη για να καλύψουμε πολλά πολιτικά στοιχεία που αφορούν την ε, λειτουργία του κράτους δικαίου. Και την Παρασκευή θα έχουμε τον τρίτο διάλογο ε, με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και την Κροατία σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών με Προεδρία του Επιτρόπου Φίλε. Εκεί οι Εξωτερικών θα εξετάσουν όλα τα συνοριακά ζητήματα και τα θέματα διέλευσης προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος και να ανεβρεθεί λύση για τα πολύ σημαντικά εκκρεμή ζητήματα που υπάρχουν για τα σύνορα αυτή τη στιγμή και θα μπορούσαν να βλάψουν την Βοσνία μετά την 1η Ιουλίου, μετά δηλαδή την ε, προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να αποφύγουμε οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια τη ένταξη αυτή για τη Βοσνία Ζεγοβίνη θα προτείνουμε σχετική διατύπωση στη κυρία Πάκ για να λάβει υπόψη και την έκβαση αυτής της συνεδρίασης. Την ε, προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και την ε, πρόταση για την έναρξη διαλόγου για θέματα παιδείας. Συμφωνούμε ότι η εκπαίδευση είναι νευραλγικό θέμα και θα πρέπει να επισημανθεί στις συζητήσεις μας με τη Βοσνία Ριζεγοβίνη και πολύ σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα το Μάιο, θα ξεκινήσουμε και ένα νέο διάλογο με ομάδα εργασία ε, της διεθνούς κοινότητας για θέματα παιδείας. Και μάλιστα υπάρχουν πολλοί αρμόδιοι στην Βοσνία Ζεγοβίνη Υπουργοί για θέματα εκπαίδευσης. Ευχαριστώ. Η κυρία Πακ θέλει το λόγο οπωσδήποτε. Βεβαίως θα περιλάβω στο κείμενο και ορισμένες θετικέ παρατηρήσεις. Αγαπητέ Ρούτσεκ, έχω και θετικά πράγματα, δεν λέω μόνο κριτικά. Μόνο στην προφορική μου εδώ τοποθέτηση εξέφρασα κάπως την απογοήτευσή μου. Αλλά ένα θέμα είναι σημαντικό. Η επιστροφή των προσφύγων. Υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν δωρητέ οι οποίοι προσφέρουν χρήματα για την επιστροφή των προσφύγων. Πρέπει να φροντίσουμε με κάθε μέσον να μην χαθούν τα χρήματα αυτά αυτοί οι οποίοι τα χρειάζονται σε αυτούς να καταλήξουν. Να υπάρξει δηλαδή ε, ας πούμε παροχή ρεύματο και νερού ε, για τις κατοικίες των προσφύγων. Κάτι το οποίο δεν γίνεται για παράδειγμα στην ε, Ρεπούμπλικα Σέρψκα. Και η μόνη χώρα των Βαλκανίων όπου δεν μπορούν να μεταβούν οι πολίτες του Κωσόβου είναι η Βοσνία Ριζεγοβίνη. Ακόμα και στη Σερβία μπορούν να πάνε αλλά όχι στη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την προθεσμία για τις τροπολογίες, που είναι 25 Φεβρουαρίου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά και να ευχαριστήσω εκ μέρους των μελών της Επιτροπής τον ε, Αντιπρόεδρο της Ελλαδικής Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών και Εμπορίου, τον κύριο Γκίλαμορ, που ε, ήρθε στην Επιτροπή μας αμέσως μετά τη λήξη του Συμβουλίου ε, Υπουργών Εξωτερικών. Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να σας ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του Προέδρου μας, του κυρίου Μπροκ, που έχει πολύ σημαντικά θέματα στην Γερμανία, γι' αυτό και δεν μπόρεσε να προεδρεύσει σήμερα στη συνεδρίαση της ΑΦΕΤ. Ε, από ό,τι ξέρω, το θεματολόγιο του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου ήταν πολύ φορτωμένη. Εξετάστηκε την κατάσταση στο Μαλί. Ελπίζουμε να αποσταλεί ε, επιτέλους η αντιπροσωπεία μας και η αποστολή μας για την ενίσχυση του στρατού του Μαλί. Και μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τι είπαν οι υπουργοί για την κατάσταση στην Ουκρανία, την τη Γεωργία και την Μολδαβία όπου η φιλοευρωπαϊκή συμμαχία αντιμετωπίζει κρίση. Εξετάστηκε και η κατάσταση στο Ιράκ, χώρα με την οποία συνήψαμε μια πολύ σημαντική συμφωνία συνεργασίας. Μας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις και στις γειτονικέ μας χώρες και νοτίως αλλά και στη Συρία και επίσης η, η, διαδικασία στην Αγγής Ανατολή μετά την έκβαση των ε, εκλογών στο Ισραήλ ιδιαίτερα. Πολύ λοιπόν ε, με στη ε, ημερή σε διάταξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως φαντάζεστε έχουμε διαβάσει τα συμπεράσματα. Περιμένουμε όμως από εσά να μας ενημερώσετε για το τι διεμειφθεί στη συνάντηση αυτή. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στον κύριο Μπρόκ να του το διαβιβάσετε σας παρακαλώ Κατανοώ ότι έχει εσωτερικά πολιτικά ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει. Το Συμβούλιο τελείωσε μία ώρα πριν περίπου, συνεδριάζαμε από τις 9.30 το πρωί και είχαμε πολύ, μια πολύ μεγάλη ημέρα με μακρόπνες συζητήσεις και χαίρομαι που βρίσκομαι ενώπιον της ΑΦΕΤ για να σας μιλήσω για την έκβαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών. Λάβαμε υπόψη την πολιτική κατάσταση στο Μαλί μετά από την έγκριση του οδικού χάρτη από τις αρχές του Μαλί και τη συνάντηση της 5ης Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες υπό την Προεδρία της ΥΠΑ εκπροσώπου της Λέδης Άστον η διαδικασία εκπαίδευσης έχει αρχίσει μετά από την ε, λήξη των ε, διαδικασιών. Το Συμβούλιο έφτασε σε συμπεράσματα με βάση την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον οδικό χάρτη εν ώψη των εκλογών αργότερα κατά το τρέχον έτος και την ανάγκη ε, του ελέγχου των στρατιωτικών δυνάμεων από πολιτικές δυνάμεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την βοήθεια και την αρρωγή που ανακοίνωσε ο Επίτροπος Πίμπαλξ στις 12 Φεβρουαρίου στο Δουβλίνο. Η απάντησή μας ως προς την κρίση στο Μαλί θα πρέπει να ε, ε, λάβει υπόψη ΚΕΠΑ, τα, τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της ε, ΚΕΠΑ με τα 50 50 ε, εκατομμύρια ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και τα 152 εκατομμύρια τα οποία είχαν δοθεί για να αντιμετωπιστεί η, χρήση, η κρίση στο Σαχέλ και τα 250 εκατομμύρια που προβλέπονται μέσα στα πλαίσια της γενικότερης ανθρωπιστικής βοήθειας, μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Το ανατολικό ε, μέτωπο ήταν ε, επίσης ένα σημαντικό ε, μέτωπο. Μιλήσαμε λοιπόν για την ανατολική εταιρική σχέση μετά τη συνάντηση στο Βίλνιους το Νοέμβριο. Θεωρήσαμε ότι με την Γεωργία, Ουκρανία, Αρμενία ε, και Μολδαβία θα πρέπει να προωθούν σχέσεις ε, ελεύθερου εμπορίου αυτό αφορά και το Αζερβαϊτζάν. Θεωρήσαμε ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να οδηγήσει στη διάσκεψη ε, κορυφής. Ο Επίτροπος ε, Φούλε μας μίλησε για τον διάλογο ανατολικής εταιρικής σχέσης στην Τυφλίδα που προωθήθηκε στην ε, Τυφλίδα την προηγούμενη εβδομάδα. Μετά από ανταλλαγή απόψεων και τη συνάντηση του Βίλνιους λάβαμε υπόψη και το, τα φόρα της κοινωνίας των πολιτών. Και αυτό καταδεικνύει τη σημασία που προσδίδουμε σε μια ανοιχτή διαδικασία εν ώψη της διάσκεψης κορυφής. Επίσης, μιλήσαμε για την ανατολική εταιρική σχέση γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες αυτές θα ορίσουν το μέγεθος της συνεργασίας και με τις μεταρρυθμίσεις θα ευεργετηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτάνοντας ε, στη συνάντηση του Βίλνιους θα φτάσουμε σε αυτά αποτελέσματα. Ως προς τη Συρία θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε με τα περιοριστικά μέτρα για τρεις μήνες επιπλέον έτσι ώστε να δοθεί και η τεχνική βοήθεια και η προστασία των αμάχων έγινε ανταλλαγή απόψεων για το πώς μπορούμε να ε, προωθήσουμε τη δράση της αντιπολίτευσης για να βρεθεί μια πολιτική λύση και ανθρωπιστική βοήθεια, να χορηγηθεί ανθρωπιστική βοήθεια. Δώσαμε μεγάλη σημασία στην εξέβρεση μιας πολιτικής λύσης, λαμβάνοντας υπόψη και τη συμμαχία της αντιπολίτευσης για να καταπολεμήσει το καθεστώς του Ασάντ θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το ανθρωπιστικό σκέλος και ε, μόνο στο Συμβούλιο του Μαρτίου Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών θα προωθηθεί και η δραστηριότητα του ειδικού εκπροσώπου του κυρίου Μπραχίνη. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουν οι άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών στη μέση Ανατολή γνωρίζετε ποια είναι η θέση μας για την έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων και αυτό το τονίσαμε πολλές φορές. Θέλουμε μία ε, λύση που να βασίζεται σε, στα αποτελέσματα και ε, λεγόμενα του Προέδρου Ομπάμα. Η ύπατη εκπρόσωπος ε, ε, αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κέρι. Ως προς το Ιράκ είναι ιδιαίτερα βάλωτο λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνοτικές μειονότητες και εντάσεις. Αποφασίστηκε από την ύπατη εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για να προωθήσουμε την ε, ε, σταθερότητα με βάση τη συνεργασία, τη Συμφωνία Συνεργασίας Ιράκ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό αφορά και τις χώρες του Περσικού κόλπου, Τουρκία και άλλες γείτονες χώρες. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, χρηστή διακυβέρνηση μέσα στα πλαίσια των 20 εκατομμυρίων που έχουν χορηγηθεί. Ο Επίτροπος Πίμπαλξ αναφέρθηκε στα ζητήματα ασφαλείας ε, μέσα στα πλαίσια χορήγησης βοηθείας στο Ιράκ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Επίσης, ε, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να καταπολεμηθούν ε, οι πυρηνικές δοκιμές και να ε, λάβουμε υπόψη και να απαγορευτούν οι πυρηνικές δοκιμές στη Βόρεια Κορέα. Θα πρέπει λοιπόν να ε, σταματήσει το νέο βαλιστικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας. Επίσης, ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, το, ε, η διάσκεψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, των Ηνωμένων Εθνών θεώρησαν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα περιοδικής αναθεώρησης. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει μία θεματική προσέγγιση μέσα στα πλαίσια του 2013. Άρα μας απασχόλησε η Σρι Λάνκα, το Μαλί, το Μιανμάρ, η Λευκορωσία, η Βόρειος Κορέα και θεωρήσαμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις με βάση τον ε, σεξουαλικό προσανατολισμό. Ως προς τη Ζιμπάμπουε φτάσαμε σε συμπεράσματα θεωρώντας ότι θα πρέπει να ανανεωθούν τα περιοριστικά μέτρα ε, ως πρόσωπα και φορείς. Επίσης ε, θεωρήσαμε και ενθαρρύναμε τα πολιτικά κόμματα να οικοδομήσουν μέτρα εμπιστοσύνης μέσα στα πλαίσια του νέου οδικού χάρτη. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, αλλά η προσέγγιση μας θα ε, θα εξαρτηθεί από την πολιτική πρόοδο που θα επιτευχθεί σε αυτή τη χώρα. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ενδεχόμενες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα... Δίνω το λόγο στους συναδέλφους για παρεμβάσεις. Και πρώτα στον κύριο Σαλαφράνκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Eh. Και ευχαριστώ και τον ε, Αντιπρόεδρο. Νομίζω ότι ήταν το, πιο, ε, το, το, ταχύτερο συμβούλιο που γνωρίσαμε στην ιστορία των, των, ε, των συνεδριάσεων του των Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών. Σε σχέση με τα συμπεράσματά σας, ε, για τη Συρία, σχετικά με τη Συρία, πέρα από τις γνωστές αναφορές του Αραβικού Συνδέσμου και του ειδικού αποσταλμένου στη Συρία από τα Ηνωμένα Έθνη και πέρα από τις παρενέσεις που ε, δίδονται μέσα στα πλαίσια του Συμβουλίου Ασφαλείας έτσι ώστε η Κίνα και η Ρωσία να αναλάβουν τις ευθύνες τους θεωρείται ότι θα πρέπει να αχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι πέτοι έτσι ώστε να αποδοθούν ευθύνες και έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια σωστή μετάβαση και αλλαγή καθεστώτος. Ως προς τις παρενέσεις σας για τη Βόρειο ε, Κορέα και την, το ψήφισμα 2084 υπάρχει μία σειρά κυρώσεων, ξεχωριστών, αυτονόμων κυρώσεων. Μπορείτε να μας ε, πείτε πώς ακριβώς έχουν. Και τέλος, σε σχέση με την αποστολή στο Μαλί, θα τύχει υποστήριξη θα, θα, θα τύχει υποστήριξης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή προβλέπεται μία αποστολή ε, στην πρωτεύουσα Μπαμάκο. Τι πιστεύετε ότι θα αποδώσει αυτή η αποστολή. Πιστεύετε ότι πρόκειται για ετοιμοπόλεμη μονάδα. Μπορείτε να μας πείτε κατά πόσο αποτιμήσατε τις συνθήκες ε, ασφάλειας αυτής της αποστολής έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τελεί υπό απόλυτη ασφάλεια αυτή η αποστολή ταχείας ε, επέμβασης. Ο κύριος Ντονζόν. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ για να μας μιλήσετε άμεσα για τα αποτελέσματα του Συμβουλίου. Σε σχέση με το Μάλι, κατά την επίσκεψη του Αντιπροέδρου Μπάιντεν στο Παρίσι εδώ και δύο εβδομάδες, ανακοινώθηκε ότι η αμίσμα, αυτή η ειδική ε, δύναμη της ε, Αφρικής, δύναμη ταχείας επέμβασης, στην οποία βασιζόμαστε ιδιαίτερα στο Βόρειο Μαλί, αυτή η στρατιωτική δύναμη θα μετατραπεί σε ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι αλλάζει η εντολή, η χρηματοδότηση, η στρατιωτική συμμετοχή και η ενδεχόμενη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε περισσότερα στοιχεία για το τι θα γίνει, αυτή, τι θα γίνει με αυτή την αποστολή ε, ειρήνευσης που θα είναι μια ειρηνευτική δύναμη. Μετά ως προς τη Συρία και το εμπάργο ε, των όπλων ελέγχθη ότι αυτό το εμπάργο ελήφθη υπόψη, δηλαδή παρατάθηκε, αλλά θα πρέπει να ε, δούμε τι θα γίνει και με τους αμάχους. Τι, τι σημαίνει αυτή η τροποποίηση και τι καλύπτει επακριβώς. Σημαίνει ότι αποδυναμώνεται η θέση μας ως προς το εμπάρκο των όπλων. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Παλέτσκης. Ευχαριστώ. Κύριε Ποριέ, Μία ερώτηση για μία χώρα που είναι η γειτονική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Λευκορωσία, περίπλοκος γείτονας. Γνωρίζετε την κατάσταση στη χώρα, γνωρίζετε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, συνεχίσει τις σχέσεις ε, με τη Λευκορωσία, επιβάλλοντας όμως κάποιες κυρώσεις και επικρίνοντας ε, την, τις αρνητικές πτυχές της πολιτικής. Δύσκολη ισορροπία μεταξύ των δύο προσεγγίσεων. Ποια είναι η δική σας γνώμη για τη στάση που θα πρέπει να κρατήσουμε απέναντι στη Λευκορωσία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Άτκινς. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω κύριε Υπουργέ. Ε, είναι σημαντικό και είναι από τα από τις πιο απολαυστικές πτυχέ τη ε, δουλειά να συναντιόμαστε τόσο συχνά με υπουργού εξωτερικών. Ελπίζω να είναι το ίδιο διασκεδαστικό και για εσά. Ε, θα θέσω μια ερώτηση για ένα ζήτημα που επανέρχεται πολύ συχνά. Τη Μέση Ανατολή. Και με τι ε, ε, εκλογές του Ισραήλ που δεν έχουν αναδείξει ακόμα κυβέρνηση, έχουμε μια μοναδική ευκαιρία ώστε να ασκήσουμε μέσω Υπουργικού Συμβουλίου ε, πίεση για να επιληθεί το θέμα των επικισμών τα ε, κατεχόμενα και γενικώ να δοθεί μια λύση στην κατάσταση. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει με κάποιο διάβημα. Σκοπεύει η Προεδρία ή η η πρόσωπος να πραγματοποιήσει αυτό το διάβημα στη συγκεκριμένη στιγμή. Ένα άλλο θέμα. Μια και συμμετέχουμε στο κουαρτέτο, μια και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέρος του κουαρτέτου, δεν θα ήταν σκόπιμο να προσκαλέσουμε τον κύριο Μπλερ να έρθει στη συνεδρίασή σας και να εξηγήσει τι κάνει το κουαρτέτο, αν κάνει πραγματικά κάτι. Ευχαριστώ κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω εκ μέρους των Πρασίνων ε, τον Υπουργό στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη για τη Συρία. Μπορεί να μην άκουσα όλα όσα είπα, ε, αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έγινε ε, λόγος για άρση των αστρατικών κυρώσεων προς τη Συρία. Η ε, παροχή όπλων προς τους ε, ανδάρτες. Τι συζήτηση έγινε για το θέμα αυτό, ποιες χώρες ήταν υπέρ. Ε, τελικά δεν έληφθη απόφαση. Υπήρξε απόφαση να μην αρθούν οι κυρώσεις, αλλά μπορείτε να μας πείτε πώς διεξήχθη η συζήτηση. Δεύτερο θέμα, Ουκρανία η κατάσταση είναι στάσιμη. Υπάρχει δυνατότητα πρόοδου. Πιστεύετε ότι θα σημειωθεί πρόοδο στο μέλλον. Προ το παρόν υπάρχει μία αποτελμάτωση πάντω. Συζητήθηκε καθόλου το θέμα αυτό. Υπάρχει κάποια ελπίδα να σημειωθεί πρόοδο στο εγγύ μέλλον, τις επόμενε δύο εβδομάδες ας πούμε. Ευχαριστώ και θα δώσω το λόγο να απαντήσει στις ερωτήσει και μετά να περάσουμε σε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Έχω ήδη τρεις ε, ομιλητές για το δεύτερο γύρο. Κύριος Υπουργός. Um, Ευχαριστώ. Καταρχήν, ως προς ερωτήσεις για τη Συρία. Του κύριο Σαλαφράγκα, του κύριο Ντανζόν, και της κυρίας Λούνατσεκ. Σε ό,τι αφορά τη θέση του Διεθνούς ε, Ποινικού Δικαστηρίου. Ένα από τα συμπεράσματα προέβλεπε, προέβλεπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για την εκτεταμένη και παρελειμμένη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, που ε, διαπίστωσε η Εξεταστική Επιτροπή. Ίσως ε, με βάση το καθεστώς της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ε, υποβληθούν κατηγορίες για, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Θα γίνει συζήτηση με τη Συρία και ίσως παραπενθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστηρίο όπως αναφέρεται στην επιστολή της 14ης Ιανουαρίου 2013 προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Και επίσης γίνεται έκκληση να προσαχθούν οι αυτοργοί ε, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Υπάρχει δηλαδή στα συμπεράσματα άμεση μνήα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε σχέση με τη Συρία. Σε ό,τι αφορά τώρα τις κυρώσεις. Οι αποφάσεις καταρχήν ενέκριναν την παράταση για ένα ακόμη τρίμηνο των υπαρχουσών κυρώσεων προς τη Σύρια. Το ζήτημα που προέκυψε δεν αφορούσε τόσο την άρση του εμπάργου όπλων, γιατί δεν πρόκειται να αρθεί το εμπάργο των όπλων. Ισχύει, εξακολουθεί να ισχύει το εμπάργο των όπλων. Αυτό που διευκρινίστηκε αφορά τη, τις διατάξεις των κυρώσεων που προβλέπουν τη χρήση μη θανατηφόρων στρατητικών εξοπλισμών και την παροχή τεχνικής αρρωγής και περαιτέρω υποστήριξης των αμάχων. Και στη συζήτηση έγινε διευκρινήση ότι μη θανατηφόρα όπλα και θα, στρατιωτικός εξοπλισμός και τεχνική ε, υποστήριξη ε, εφόσον δεν έχουν, αφορά θανατηφόρα μέσα μπορεί να παρα, παρασχεθεί με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των αμάχων. Αυτό όμως δεν σημαίνει όπως λένε τα συμπεράσματα, ότι θα έρθει το εμπάρκο των όπλων ούτε κατά διάνοια δεν εξετάστηκε η πιθανότητα άρσης του εμπάργου όπλων στη Συρία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Μαλί. Έγινε μία ενημέρωση από κάποιες χώρες μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάσταση ασφάλειας ό,τι αφορά το Μαλί και ιδιαίτερα την ανθρωπιστική κατάσταση. Η γαλλική στρατιωτική επιχείρηση στο Μαλί με πάνω από 4.000 στρατιώτες συνεχίζεται με την υποστήριξη κάποιων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών φορέων. Και μάλιστα ε, έχουμε και την ΦΙΣΜΑ που περιλαμβάνει 2.000 στρατιώτες από το Τσάτ και που μένουν εκτός ε, της επιχειρησιακής ευέλειας ε, της ΦΥΣΜΑ. Πάντως ε, τα βόρεια του Μαλή απελευθερώθηκαν από τρομοκρατικά στοιχεία χάρη στην ε, στην Ποκτού, Γκάο και Κιτάτ και μάλιστα μερικοί χρησιμοποίησαν ε, ανταρτοπόλεμο μερικοί τρομοκράτες αλλά έχουν απελευθερωθεί πια τα βόρεια χάρη στη συνεργασία του στρατού του Μαλή με την με τις γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις. Σε ό,τι αφορά την Ανατολική Γειτονία, κύριε Παλέτσκης, και κυρία Λούνατσεκ, αναφερθήκατε στην Λευκορωσία και την Ουκρανία. Το σημαντικό σήμερα είναι ότι έγινε συζήτηση πολύ πριν την Υπουργική Διάσκεψη του Ιουλίου και την Υπουργική Διάσκεψη του Νοεμβρίου. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων μεριμνά καταρχήν για την σωστή προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής της Τυφλίδας και μας ενδιαφέρει επίσης στο εγγύς μέλλον να δώσουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα στην ε, Ανατολική Γειτονία και στις χώρες που περιλαμβάνει αυτή. Και αυτό αφορά και τις ε, ενταξιακές τους βλέψεις, πώς βλέπουν ε, το μέλλον τους, τι κατεύθυνση θα ακολουθήσουν ποια είναι η προοπτική τους για την Ένωση, τι γίνεται με τις ε, συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, θέματα δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτος δικαίου και η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα της Ανατολικής Γειτονίας. Δεν ισχύει μια ενιαία κατάσταση σε όλες τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας, Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Η κατάσταση διαφέρει, επαναλαμβάνω, από χώρα σε χώρα Γι' αυτό και το θέμα αυτό θα απασχολήσει και θα απασχολεί τακτικά το Συμβουλίο Εξωτερικών Υποθέσεων. Κύριε Άτκινς, ε, ρωτήσατε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Στη συζήτηση που είχαμε στο γεύμα για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, είπαμε ότι πραγματικά ανοίγεται ένα παράθυρο ευκαιρία και σίγουρα αμέσω μετά τι προεδρικέ εκλογέ των Ηνωμένων Πολιτειών και μετά τι ε, ε, Ισραηλινές εκλογέ, θεωρήσαμε ότι θα δημιουργηθεί μια ευκαιρία για να σημειωθεί πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία τη Μέσης Ανατολή. Και μάλιστα μα ενθάρρυναν ιδιαίτερα τα σχόλια του νέου Υπουργού Εξωτερικών τον ΙΠΑ, του Τζον Κέρι, για το ενδιαφέρον που δείχνει για την ειρηνευτική αυτή διαδικασία και ο πρόεδρος Ομπάμα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ισραήλ, κατά πάσα πιθανότητα το Μάρτιο ή εκεί γύρω. Οπότε υπάρχει μια ευκαιρία να δραστηριοποιηθεί έντονα η Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεργαστεί και με άλλους ε, παγκόσμιους φορείς ώστε να προωθήσει μία διευθέτηση, μία συμφωνία στη Μέση Ανατολή. Να δοθεί μία όθηση στο διάλογο. Θα πρέπει βέβαια να δούμε και το ρόλο της τετραμερούς διάσκεψης, του κουαρτέτου και πώς εντάσσεται ο ρόλος αυτής της διάσκεψης τετραμερούς ε, στη συζήτηση που θα διεξαχθεί. Δεν ε, εξετάσαμε τη δυνατότητα να προσκαλέσουμε τον κύριο Μπλερ σε ένα Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχουμε στο κατάλογο τον καλεσμένο μας τον δόκτωρα Αμπραχήμι, μάλλον στο Συμβούλιο του Μαρτίου, για να συζητήσουμε την κατάσταση στη Συρία. Αλλά δεν έχουμε εξετάσει ακόμη την πρόσκληση του Τόνι Μπλερ. Αν ξέχασα κάτι, παρακαλώ να μου το υπενθυμίσετε. Ευχαριστώ. Δεύτερος γύρος, ο κύριος Πέτερινγκ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών. Δεν σας ζηλεύουμε. Στα καθήκοντά σας ο κόσμος είναι μεγάλος και τα προβλήματα επίσης μεγάλα και ποικίλα. Μία ερώτηση για το Μαλί. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να ευγνωμονούμε τον πρόεδρο της Γαλλίας που ανέλαβε δράση στο Μαλί. Δεν νομίζετε όμως ότι τέτοια στρατιωτική δράση θα έπρεπε να είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις εμπειρίες του Μαλή. Έχετε δει πέσα άλλωστε το Γενικό Γραμματέα της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων, τον Πιερ Βιμό. Μήπως υπάρχουν σκέψεις ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν κάποιες στρατιωτικές δομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε στο μέλλον τέτοιες προκλήσεις να μπορούν να αντιμετωπίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τέτοια, όπως αυτές δηλαδή του Μαλή και που όπως είπα ευτυχώς ανέλαβε στρατιωτική δράση ο, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας αν και θα έπρεπε να είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η άποψή σας. Ο πρόεδρος ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Ρότσεκ. Ευχαριστώ και εγώ. Να μείνουμε στη Μέση Ανατολή. Είπατε κύριε Υπουργέ ότι θα πρέπει να δράσουμε, να είμαστε proactive εφόσον ανοίγεται κάποια ευκαιρία Τώρα αυτό ακόμα περισσότερο με τη δεύτερη θητεία του Πρόεδρου Ομπάμα. Να σας ρωτήσω για την Εσμπολάχ. Διότι υφιστάμεθα πιέσεις από τους Αμερικανούς και τους Αμερικανούς βουλευτές του Κογκρέσου να βάλουμε την Εσμπολά στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων μετά από κάποια πρώτα συμπεράσματα των βουλγαρικών αρχών σχετικά με τους φόνους του Μπουργκάς συζητήθηκε το θέμα αυτό και πώς βλέπουμε ως Ένωση την Εσμπολάχ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ είμαι κύριε Υπουργέ. Ήδη με κάλυψε η κυρία Λούνατσεκ για την Ουκρανία και την Ανατολική γειτονία. Βλέπετε να διαγράφεται πιθανότητα υπογραφής της DCFTA, δηλαδή της ε, Συμφωνίας Συνδέσεως, εφόσον δεν έχουν γίνει παρκής μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία. Χαίρομαι για την απόφαση του Συμβουλίου για την Ζιμπάμπουε. Εγώ έχω διαρκείς επαφές με την οργάνωση Justice for Zimbabwe, δικαιοσύνη για τη Ζιμπάμπουε, για την αποζημίωση αγροτών από το καθεστώς Μουγκάμπε. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι θα μελετηθεί το θέμα αυτό και θα ληφθεί υπόψη στο μέλλον όταν θα αναθεωρηθεί το καθεστώς των απαραίτητων κυρώσεων για τη χώρα αυτή. Για την Εσμπολάχ, που και εγώ ήθελα να θέσω το ίδιο θέμα, μετά από τις θηριωδίες αυτές στην Βουλγαρία, η Ιρλανδική κυβέρνηση ήταν αυτή που ήταν αντίθετη συνήθως να περιγραφεί η Εσμπολάχ ως τρομοκρατική οργάνωση. Με την αιτιολογία που ίσως μπορείτε να μας εξηγήσετε, ότι υπάρχει μια διάκριση μεταξύ της στρατιωτικής πτέρυγας που ε, είναι ε, θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση και του πολιτικού τμήματος που δεν είναι. Ενώ η ίδια η Εσμπολάχ δεν κάνει τέτοια διάκριση, θεωρεί ότι είναι μια ενιαία οργάνωση. Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε λοιπόν την θέση της κυβερνήσεώς σας και γιατί η Εσμπολάχ δεν έχει ακόμα μπει στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Άλλος κανείς. Καλά λοιπόν, θα παρακαλέσω τον Υπουργό να απαντήσει. Με συγχωρείτε, λέει ο Πρόεδρος. Follow-up ερώτηση του κ. Τανζάν. Επανέρχομαι στο θέμα του Μαλή και την μετατροπή των Αφρικανικών δυνάμεων, άφισμα, σε την υπαγωγή τους δηλαδή στα Ηνωμένα Έθνη, την μετατροπή τους αν θέλετε σε αποστολή των Ηνωμένων Εθνών. Πού βρισκόμαστε εκεί. Κύριε Υπουργέ. Okay, let me take, um... Ας αρχίσουμε πρώτα από το Μαλί και να πω εξ αρχής ίσως μάλιστα έπρεπε να το είχα πει και πριν απαντώντας, ότι έχουν γίνει σημαντικές προετοιμασίες για την εκπαιδευτική αποστολή της ε, εκπαίδευση των δυνάμεων εκεί με Γάλλο διοικητή και να αρχίσει η εκπαίδευση των ε, μαλιακών δυνάμεων αρχές Απριλίου με συμμετοχή 200 εκπαιδευτών και μαζί με την ε, δημιουργία επιτελείου στην Μπαμάκο με υποστήριξη επιμελητίας με ένα συνολικό αριθμό προσωπικού περίπου 500 ατόμων και με επιτελείο στο Νουρικόρο που είναι περίπου 500 χιλιόμετρα από το Μπαμάκο. Πάντως δεν έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία αυτή και προωθείται τώρα όσο γίνεται ταχύτερα για να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν και τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και ώστε να μην χαθεί χρόνος έτσι ώστε να μπορέσει η στρατηγική εκπαίδευση να αρχίσει αμέσως. Για το εάν η ανταπόκριση μας την κατάσταση που διαμορφώθηκε στο Μαλί θα πρέπει να είναι η ευθύνη, η καθήκον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή μεμονωμένων χωρών μελών που ενδεχομένως θα αναλάβουν την ευθύνη αυτή. Ένας από τους παράγοντες που πρέπει να ληφθεί υπόψη νομίζω είναι και η ευνίδια εξέλιξη της κρίσης αυτής και κατά κάποιο τρόπο η Γαλλία ήταν σε θέση να παρέμβει ταχαίως λόγω της στάθμευσης δυνάμεών της στο Τσάντ, την Σενεγάλη και την ακτή του Ελεφαντοστού. Και το θέμα των μελλοντικών ενδεχομένω ευρωπαϊκών δομών στον χώρο της άμυνας είναι βέβαια ευρύτερη συζήτηση. Στο Μάλι βέβαια, μάλλον το Μάλι και η περίπτωση του Μάλι και η ανταπόκριση που δόθηκε στο Μάλι είναι ένα θέμα το οποίο συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά βέβαια πρέπει να κριθεί αυτοδύναμα. Ελπίζω ότι με κάποιο τρόπο απάντησα στην ερώτηση σας κυρία Πέτερη. Είναι ευρύτερο θέμα, όπως είπα, και αυτό το ευρύτερο θέμα μάλλον πρέπει να γίνει αντικείμενο μακροσκελέστερης συζήτησης από ότι θα μπορούσε να χωρέσει σε τούτη εδώ την συζήτησή μας. Σε ό,τι αφορά την Εσμπολάχ και τους φόνους του Μπουργκάς, το Συμβούλιο ενημερώθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας για τα πρώτα πορίσματα της έρευνας της επίθεσης στο Μπουργκάς. Θέμα το οποίο έθεσαν οι κύριοι Ρότσο και Τάνοκ. Έγινε δεκτό ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να ενθαρρύνει τις λιβανικές αρχές να συνεργαστούν με τη Βουλγαρία έτσι ώστε οι δράστες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους στην προσπάθεια καταπολέμησης της διεθνούς τρομοκρατίας. Εν προκειμένου η διάθεση του Πρωθυπουργού να, του να συμμετάσχει είναι καλοδεχομένη. Σε αυτή την ενημέρωση του Συμβουλίου, ο Βούργαρος υπέξ προέβηκε και σε εκτίμηση για το πού βρίσκεται η έρευνα και είπε ότι θα επανέλθει σε μελλοντική συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών εφόσον θα έχουν εξαχθεί τα συμπεράσματα και θα έχουν αντληθεί τα σχετικά διδάγματα από την έρευνα. Δεν διεξήχθη ωστόσο συζήτηση σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών σχετικά με την ε, προκήρυξη της Εσμπολάχ ή με, την, τον χαρακτηρισμό της Εσμπολάχ ως τρομοκρατικής οργανώσεως. Εγώ δεν εκπροσωπώ σήμερα την κυβέρνησή μου, απαντώ στην ερώτησή σας σχετικά με τη θέση της κυβέρνησής μου, αλλά την Προεδρία του Συμβουλίου. Αλλά νομίζω ότι πρέπει όντως να εξετάσουμε την κατάσταση στο Λίβανο. Σαφώς ο Λίβανο είναι μια χώρα που κατέχει κρίσιμη θέση στην περιοχή αυτή και ιδιαίτερα κρίσιμη στην προκείμενη περίπτωση και σε σχέση με το όσα συμβαίνουν στην Συρία. Έγινε βέβαια και κάποια οικοτολογία στον τύπο για το αν συζητήθηκε στο Συμβούλιο των Εξωτερικών. Δεν έγινε τέτοιου είδους συζήτηση. και αναμένουμε τις απόψεις του Βουλγάρου υπέξ όταν και εφόσον επανέλθει η μελλοντική συνεδρίαση. Για την Ουκρανία. Προ 15 μέρου είχαμε μια ιδιαίτερα σημαντική συνεδρίαση τα μέλη του, του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό της Ουκρανίας και η προσέγγιση αυτή που λέει περισσότερα έναντι περισσότερων δηλαδή η συζήτηση για εμπορικές συμφωνίες, για συμφωνίες συνδέσεως θα πρέπει να συνεχιστούν μόνο στη βάση που θα υπάρχει κάποια ανταπόκριση από τις χώρες της, πολιτική της πολιτικής γειτονίας περιλαμβανομένης της Ουκρανίας. Αυτή είναι η προσέγγιση που θα επιλεχθεί, που θα ληφθεί και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την μόχλευση που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως την οικονομική για να επιτύχουμε πρόοδο και ιδίως στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Αλλά αυτό πρέπει να εξισορροπηθεί, αν θέλετε, και με την εξασφάλιση αλλά και ενθάρρυνση των χωρών της Ανατολικής Γειτονίας, δίνοντάς τους μια ευρωπαϊκή προοπτική. Γιατί αν χαθεί αυτή η προοπτική, τότε το εύρος, η δυνατότητα άσκησης πυθούς αλλά και πίεση στον χώρο των ανθρώπινων δικαιωμάτων μειώνεται. Όλοι βέβαια θα θέλαμε να δούμε να γίνεται πρόοδο πολύ ταχύτερα από αυτήν που σημειώνεται τώρα. Και ασφαλώς διατηρούμε σημαντικές ανησυχίες για την κατάσταση και για την Ουκρανία αλλά και ιδίω για τη Λευκορωσία. Σε ό,τι αφορά τη Ζιμπάμπουε, αγαπητέ Τάνοκ, πάλι εδώ η απόφαση σήμερα για τις κυρώσεις κατά τη Ζιμπάμπουε ελήφθη μετά από κάποια πρόοδο που επιτελέστηκε εκεί και το Συμβούλιο ΕΠΕΞ ανταποκρίνεται στην πρόοδο που έγινε με χρήση των κυρώσεων για να ενθαρρύνουν κάποια πρόοδο, εφόσον βέβαια υπάρχει πρόοδος. Γίνεται κάποια χαλάρωση των κυρώσεων έτσι ώστε να υπάρξει κάποια επιβράβευση για την πρόοδο, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να είναι πολύ μετρημένη και να αναθεωρείται διαρκώς. Το Συμβούλιο βεβαίως θα επανέλθει στην εξέταση της κατάστασης αυτής, όπως διαγράφεται στη Ζιμπάμπουε, για τον κύριο Τανζόν, για το θέμα για το ευρύτερο θέμα δηλαδή της μεταφοράς από την άφισμα σε δύναμη των Ηνωμένων Εθνών. Είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί χρόνο, θα χρειαστεί και ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς επίσης και να δημιουργηθεί μια δύναμη με καθαρή εντολή. Είμαστε βέβαια ακόμα στην αρχή της διαδικασίας αυτής. Ο πρόεδρος του Μαλή μόλις έστειλε επιστολή στον Πανκιμούν Κιμούν δίνοντας προσφέροντας την συμφωνία του, τη συμφωνή γνώμη του δηλαδή, για να δημιουργηθεί η αποστολή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν άλλες, ερωτήσεις. Άλλες παρεμβάσεις, ερωτήσεις. Φαίνεται κύριε Υπουργέ ότι ικανοποιήσατε όλους τους βουλευτές με τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε και για την προσέλευσή σας, την τάχιστη προσέλευσή σας μετά τη λήξη, με τη λήξη του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών. Ε, αναμένουμε να σας ξαναδούμε και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και στις μελλοντικές σας δραστηριότητες.